Colleagues, good morning. Next item on the agenda is the chairman's announcements and of course that's the Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι ανακοινώσεις ε, του Προέδρου, τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών και ο διορισμός ε, των εισηγητών, ε, των συνεισηγητών, των σκιωδών εισηγητών κτλ. Όσον αφορά τους εισηγητές και τους συντάκτες, έγινε μια συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, στην, και στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για να συντονίσουμε ε, την συνεδρίαση. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα κάνουν την ε, έκθεση. Θα δούμε τώρα όμως ποιοι, ε, ποιος, ποιοι αντιπρόεδροι έχουν δουλειά και ποιοι δεν έχουν για να δούμε. Τώρα, για τα άλλα θέματα, ήταν ένα έγγραφο της Κομισιόν για την ε, τεχνολογία, την ε, εναέρια κυκλοφορία κτλ. Για ε, τεχνολογία κτλ. Στην πέμπτη έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού 2321 για την ασφάλεια στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Μία έκθεση χρειάζεται. Οι συντονιστές δεν αποφάσισαν, αλλά θα ζητήσουμε από τον, από τον κύριο Πασκουάλ να συμπε να τα συμπεριλάβει το θέματα αυτά στη δική του έκθεση για την ενέργεια ασφάλεια. Τώρα, για τα επόμενα δύο θέματα, για τους ελέγχους των αεροσκαφών και για την, τις μεταφορέ. μεταφορές, θα πούμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε ακόμα. Τώρα για τις γνωμοδοτήσεις ε, για τον, για τον Δούναβη, για την ανακοίνωση της Κομισιόν, οι συντονιστές δεν πήραν απόφαση, γιατί όπως ξέρετε η Περιφερειακή Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει ε, μετά από αυτή την ανακοίνωση. Ε, εάν η Επιτροπή, Περιφερειακή Επιτροπή κάνει κάτι, τότε θα πρέπει και εμείς να γνωμοδοτήσουμε, γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα καθαρά και αποτελεσματικά οχήματα, ε, είναι ένα έγγραφο εργασίας, τέλο πάντων, του προσωπικού, ε, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Τώρα, όσον αφορά την αναθεώρηση του χρόνου εργασίας και την εφαρμογή από πλευρά των κρατών μελών ε, της οδηγίας 88 του 2003 και όσον αφορά το έγγραφο εργασίας ε, για την εφαρμογή το, το 2000, 2007-2008 ε, του, του κανονισμού 561 όσον αφορά την, τις οδικές μεταφορές δεν είμαστε Εμεί ακόμα δεν, δεν, περιμένουμε από την άλλη επιτροπή να γνωμοδοτήσει. Δεν ξέρουμε ε, εάν θα γίνει αυτό. Γι' αυτό είπαμε να, να καταρτήσουμε 5-6 ερωτήσεις, να... τις οποίες απευθύνουμε στην Κομισιό και να στην επόμενη Επιτροπή Μεταφορών να εξασφαλίσουμε απάντηση για αυτές τις ερωτήσεις. Θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει ε, σε αυτό το τομέα, αλλά επειδή η Επιτροπή Απασχόλησης δεν κάνει γνωμοδότηση, ο μόνος τρόπος για να μάθουμε πέντε πράγματα παραπάνω είναι να ε, κάνουμε την ερώτηση στην Κομισιό. Αυτό αποφάσισε οι αποφάσισαν συντονιστέ. Τώρα για την αναθεώρηση του προπολογισμού, στις 8 Νοεμβρίου η συνεδρίαση ε, των συντονιστών ανέβαλαν την απόφαση. Εν τω μεταξύ όμως η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού ε, αποφάσισε να μην κάνει τίποτα. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας και όλα τα έγγραφα τα οποία κυκλοφορούν για το θέμα αυτό και οι συντονιστές είπαν θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή ΣΟΥ. Τώρα, για την, για την εσωτερική αγορά, η Επιτροπή για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, οι συντονιστές ε, αποφάσισαν ότι επειδή δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο και το χρονοδιάγραμμα της ΙΜΚΟ είναι πάρα πολύ στενό σε σχέση με την ανακοίνωση για την ενιαία αγορά, είπαμε ότι θα ε, υπάρχει μια επιστολή, θα στείλει ο πρόεδρος μια επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΜΚΟ και οι συντονιστές θα, μέχρι τις 31 ε, Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβάλλετε στον ε, γραμματέα της Επιτροπής μας οποιασδήποτε αλλαγές θέλετε και οποιασδήποτε προτάσεις έχετε για την επιστολή και με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά στον πιο γρήγορα με την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Εγώ Μίλησα με τον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΜΚΟ και συμφωνεί με την ε, διαδικασία και θεωρεί ότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Μεταφορών, πρέπει να έχει μια συνεισφορά σε αυτά τα οποία γίνονται. Τώρα, όσον αφορά την στρατηγική 2020, οι συντονιστές συμφώνησαν να υποβάλουν οποιασδήποτε αλλαγές ε, στην επιστολή του Προέδρου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου στις 3 η ώρα, μέχρι τις 26 συγγνώμη, Ιανουαρίου στις 3 η ώρα ε, και θέλουμε να υπάρχει μια συνεισφορά έτσι, από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες έτσι ώστε ε, να μπορούμε το Μάρτιο του 2011 στην Σύνοδο Κορυφής να συνεισφέρουμε και εμείς. Λοιπόν, μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, 3 η ώρα, θέλω τις προτάσεις σας για να μπορέσω να τις εντάξω στην επιστροφή. Τώρα, όσον αφορά την επιτροπολογία, ο αντιπρόεδρος Ρίκε πρότεινε να παρακολουθήσουμε από κοντά τα όσα συμβαίνουν με το ITS και να το συζητήσουμε στην Επιτροπή και η πράσινη μέσω της κυρίας Λίχτενμπέρκερ ζήτησε ε, την προστασία των πεζών από τα λεωφορεία. Ε, ο αντιπρόεδρο Φαντάλεν έθεσε το θέμα κάποιων διπλωμάτων οδήγηση και ο κύριος Αλκαντάλτρη, ο οποίο είναι ε, ο εισηγητήσει γενικά τα θέματα επιτροπολογία, είπε ότι θα μα κρατήσει ενήμερου. Τώρα όσον αφορά το, το θέμα που έδειξε ο αντιπρόεδρο Βαντάλε για του ε, πιλότου, τις ιδιώτε πιλότε, αν θέλετε, πιλότου ιδιωτικών αεροπλάνων, ε, ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα έχει ένα κείμενο το Φεβρουάριο να μας διαβιβάσει. Αυτό είναι θέμα, τα θέματα των ε, πιλότων ιδιωτικών αεροσκαφών που έχουν διπλώματα από την Αμερική. Αυτά θα τα συζητήσουμε το Φεβρουάριο ε, και ίσως ανταχθούν στην, ε, στους συντονιστές και θα ανταχθούν στην ημερήσια διαταξή μας τον Μάρτιο. Στα διάφορα, οι συντονιστές δέχτηκαν την, ε, υπε, την παρέτηση του κύριου Κόξ και ο κύριος Κόξ πρότεινε να αντικατασταθεί ο κύριος Κότσο από έναν άλλον συνάδελφο. Μια συζήτηση για τα θέματα αυτά αλλά η σύσταση των συντονιστών έτσι όπως είναι, είναι ο κύριος Γκάντσιαν να αντικαταστήσει τον κύριο Κότσου. Τώρα, ζητήσαμε ε, μία ε, ενημέρωση για το, τα θέματα αποδέσμευσης στον τομέα των συνδρομικών μεταφορών και ζητήσαμε να έχουμε ένα λεπτομερές ενημερωτικό σημείωμα για την αποδέσμευση των θαλάσσιων και συνδρομικών μεταφορών ε, και το κανονιστικό πλαίσιο στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στους επόμενους δύο μήνες, έτσι ώστε να είμαστε ενημερωμένοι πριν ε, αποφασίσουμε για την έκθεση κυρία Σεργία. Α, για αυτό το σημείο θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, μόλι ολοκληρώσω θα, θα δώσω το λόγο σας και σε οποιοδήποτε άλλο θέλει να πάρει το, το λόγο. Τώρα για τη χρεοκοπία αεροπορικών εταιριών, οι συντονιστέ ζητήσαμε να στείλουμε ε, μια άλλη επιστολή στον Αντιπρόεδρο Κάνας παρά την δέσμευση της Κομισιόν να υποβάλει μία πρόταση. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία πρόταση. Επομένως, η πρόθεση είναι να ζητήσουμε τον Αντιπρόεδρο, τον κ. Κάλλας, να μας πει πού είναι η πρότασή του. Οι συντονιστές επίσης ε, συμφώνησαν να καλέσουμε ε, στις 18 Φεβρουαρίου τον ε, κύριο Κάλλας να μας παρουσιάσει το πρόγραμμά του λεπτομερώς για το 2011, τι προτάσεις για κανονισμούς μπορούμε να περιμένουμε κατά τη διάρκεια του έτους. Τώρα για τον Ρήνο, το ατύχημα στο Ρήνο, είναι να θέτει το θέμα της ε, εσωτερικής ε, ε, ναυσιπλοείας και τονίζει τη σημασία του. Οι συντονιστέ ζήτησαν να στείλουμε μια επιστολή στον αντιπρόεδρο κάλας, να δούμε τι έχει γίνει έκτοτε και πότε θα είναι ελεύθερος ο Ρήνος για την ναυσιπλοεία. Τώρα για την Ροβινιέτα, ο εισηγητής, ο κ. Σαρκατράουε, στις 24 Ιανουαρίου είχε μια συνάντηση με την Ουγγρική Προεδρία. Ε, αν το Συμβούλιο μας ενημερώσει εγκαίρως για την σύνοδο του, του... του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, έχουμε τέσσερις μήνες στη διάθεσή μας για να δράσουμε. Κάποιοι σέβονται τις, προ, ε, δεσμεύσεις ε, του, των συνθηκών, άλλες όχι. Αλλά τέλος πάντων μας πιέζει ο χρόνος, έχουμε μονάχα τέσσερις μήνες στη διάθεσή μας. Ο εισηγητές ε, θα συναντήσει τον, τους κοιόδους εισηγητές για να... συμφωνήσουμε για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την διαδεύτερη ανάγνωση με την Ουγγρική Προεδρία και στις και αυτές είναι οι ανακοινώσεις μου τώρα, ολοκληρώθηκαν. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ ζήτησε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Για τη σύντομη μελέτη για τα θέματα αποδέσμευσης. Αν θυμάμαι καλά, συμφωνήσαμε να μιλήσουμε και για την πραγματική, το πραγματικό άνοιγμα της αγοράς. Είπατε ότι είναι η αποδέσμευση μετά την θέση των ρυθμιστών, αν θέλετε, και το τρίτον είναι πώς πραγματικά θα ανοίξει η αγορά. Δηλαδή ή πόσο πραγματικά έχει ήδη ανοίξει η αγορά. Υπάρχει επιτυχία, υπάρχει μεταφορά από ιδιωτικές ε, ε ξένες εταιρείες στο δίκτυο. Και αυτό θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Κοιτάξτε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Όντως πρέπει να το σημειώσουμε. Να το δούμε. Άλλος θα ήθελε το λόγο για τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Αν όχι μπορεί, μπορούμε να, το τη συμφωνήσουμε. Οκ. Okay. Next is the votes. Πάμε στις ψηφοφορίες. Έχετε όλη την κάρτα, την κάρτα σας. Ωραία. Για να κάνω μια δοκιμή, εν περιπτώσει, για να δούμε τι, τι, ψάρια θα πιάσουμε αυτή τη βδομάδα. Ωραία λοιπόν. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Okay. This will be a complete shock to you. Guess who's two over. <laughs> The EPP. Λοιπόν, και τι γίνεται, ποιος έχει δύο ψήφους παραπάνω, το ΕΛΚ, ο συνήθως. Hey. Ωραία, φροντίστε να το ρυθμίσετε. Εμεί προχωρούμε με τη ψηφοφορία. Κοιτάξτε. Λοιπόν, υπάρχει κανείς που δεν έχει την κάρτα του. Όχι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με την με τις ενα... να αρχίσουμε τις εναέριες μεταφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Βραζιλίας. Ε, ψηφίζουμε. As everybody voted? The vote is... Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. used to this machine. So is that 38 in favour, none against, no abstentions? 38 υπέρ, κανείς κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια κυρία Τικάου, είστε η ροίδα της Βραζιλίας. Προχωρούμε. η συγγήτρια κυρία Σαναλόβα για την ε, για τις μηχανές για τους κινητήρες υπέρ κατά για την πρώτη τροπολογία απορρίπτεται σε 5 και 8 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές Α, να το ελέγξουμε ένα λεπτό. Είναι οι τροπολογίες 5 και 8, ε, του κυρίου Ρικέ. Ψηφίζουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά... Πάλι το ΕΛΚ. Ένα επιπλέον, μία ψήφος επιπλέον. Ωραία. Πέρα στις ψηφοφορίες. 20 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 4 και 6 καταπίπτουν. 3 και 7 καταπίπτουν επίσης. Πάμε κατευθείαν στην τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα προσπαθήσω μην χειροκροτήσω. Προχωρούμε. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν κλαίω τώρα. Δεκατέσσερα. 14 14 και 15 πάνε μαζί, αλλά υπάρχει μια προφορική τροπολογία Μαρσίνκεβιτς που την έχετε νομίζω είναι κανείς αντίθετος με την προφορική τροπολογία όχι, ωραία λοιπόν 14-15 υπέρ κατά αποχές για να το επαληθεύσουμε τροπολογίες 14-15 μαζί με τις προφορικές τροπολογίες παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες 21 υπέρ 18 κατά εγκρίνονται 16 με μια προφορική τροπολογία αντίρρηση όχι ωραία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία παρακαλώ ψηφίστε ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας 35 υπέρ 4 κατά καμία αποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Next item on the agenda is the policy challenges. Επόμενο θέμα, οι προκλήσεις, πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομική πόρη για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Δική μου έκθεση. Τροπολογία 1. Νομίζω ότι η τέσσερα απεσήρθη. Μέρος της τέσσερα απεσήρθη. Το δεύτερο μέρος απεσήρθη. Αυτό που λέει ειδικό προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Λοιπόν, για το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μέρος της τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Πρώτο μέρος υπενθυμίζει και τα λοιπά. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, όπως ορίζεται στους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ, κατά, αποχές. Να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 1, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες λοιπόν 18 υπέρ 20 κατά απορρίπτεται Τροπολογία 2 Αγιάλα Σέντερ υπέρ Κατά Αποχές εγκρίνεται Η 3 καταπίπτει 5 υπέρ Κατά Αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 κόζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 απεσύρθη 10 ζήλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική λύση α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 13 τώρα καλύπτεται 14 κόζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 με την προφορική τροπολογία συμφωνείτε με αυτήν ωραία για τη 15 τώρα υπέρ κατά αποχές να το ε, παληθεύσουμε παρακαλώ η 15 με την προφορική τροπολογία ψηφίστε του κυρίου Τεξέιρα ψηφίσατε Ωραία. Πέρα τη ψηφοφορία. 19 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 της κυρίας Τικάου, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές να το ελέγξουμε αυτό 17. Ψηφίστε. πέρας της ψηφοφορίας 25 υπέρ 14 κατά εγκρίνεται συμβασμός δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αντε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβασμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 καλύπτεται από το συμβιβασμό Πάμε στην 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. My advice is that we should vote amendment 27. Πρέπει να ψηφίσουμε την 27. Λέει όμως εδώ κατά πίπτη αν εγκριθεί ο συμβιβασμός Β. Εγώ λέω να ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Amendment 28 Vote is open. Ωραία. 28 ξανά. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. 17 υπέρ 21 κατά έχετε δίκιο απορρίπτεται 29 Ντάντιν με προφορική τροπολογία είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας όχι υπέρ της 29 κατά αποχές να το υπαλληθέσουμε νομίζω ότι απορρίπτεται 29 λοιπόν Ντάντιν υπέρ ε ψηφίστε συγγνώμη Πέρας της ψηφοφορία. 16 υπέρ 22 κατά απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 Ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπογραμμίζει ότι τα σχέδια μεταφορών και τα λοιπά. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. 34. Θα σα υπενθυμίσω ότι εδώ ψηφίζουμε με βάση το αγγλικό κείμενο, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το γερμανικό κείμενο. Ε? Λοιπόν, ψηφίζουμε για το... με το αγγλικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Πάλι με βάση το αγγλικό κείμενο Α, συγγνώμη, ξέχασα τη 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 το αγγλικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 πάλι η ψηφοφορία σε τμήματα να διαγραφεί η λέξη dramatically. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Το dramatically διαγράφεται λοιπόν. Φαντάζομαι ότι το υπόλοιπο κείμενο βρίσκει σύμφωνος. Λοιπόν, για το υπόλοιπο κείμενο χωρίς το δραματικά, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται το η 40 απεσύρθη 41 υπέρ α με συγχωρείτε ο συμβιβασμός Γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο συμβιβασμός Γ λοιπόν 41 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 απεσύρθη 43 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 απεσύρθη 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 με μια τροπο, προφορική τροπολογία έχει κάνει ένσταση για την προφορική τροπολογία όχι ωραία όλο μαζί λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η τελική ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ As everybody voted Πέρα is ψηφοφορία. 34 υπέρ, 0 κατά, 3 αποχές. Οπότε εγκρίνεται, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Λίχτενμπέργκερ, ζητώ συγγνώμη. Ήθελα να ψηφίσω υπέρ και όχι να απόσχω, αλλά δεν πρόλαβα. Ε, είχαμε πια στην κουβεντούλα εδώ, γι' αυτό. I have got Έχω τόσα χαρτιά εδώ πέρα πάνω που δεν μπορώ να βρω την έκθεση του κυρίου Κόλιτσεκ για την πολιτική συνοχής. Τροπολογία 1. Φλάσακ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. δύο Απεσύρθη. Προφορική τροπολογία τώρα για την παράγραφο 2α νέα του κυρίου Λιμπεράτσκι. Έχει κάνει αντίρρηση. Αν όχι, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα μέχρι το European Transport. Για το πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό. Οπότε η τρία καταπίπτει. Πέντε τώρα υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά πέντε Πέρα στις ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 6. Κυρία Τικάου, προστίκη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7. Ήταλα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι οκτώ είναι σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα μέχρι την ε, οικοαποτελεσματική μεταφορά. Για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 με την προφορική τροπολογία του κυρίου Ρικέ Υποθέτω δεν υπάρχει ένσταση για αυτή. Για το σύνολο, λοιπόν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 ως εκ τούτου καταπίπτει, 15 υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία. 19 υπέρ, 19 κατά. Ισοπαλία απορρίπτεται. 16. Ήταλα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Τικάου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Φλάσακ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 19 τικάου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία everybody voted? Ψηφίσατε όλοι Ένα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τους πράσινους ε. Τέλος πάντων λοιπόν πέρα στις ψηφοφορίες. 35 υπέρ, κανείς κατά, τρεις αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κόλιτσεκ, διαβιβάστε τα. Ευχαριστούμε συνάδελφοι, νομίζω ότι κλείσαμε με τις ψηφοφορίες. Προχωρούμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Τικάου για την εφαρμογή GNSS. Σίλβια, έχει το λόγο. Από εκεί και πέρα αυτοί που αποχωρούν ας αποχωρήσουν ήσυχα παρακαλώ. Η κυρία Τικάο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση, η σημερινή, αφορά το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης, GNSS. Στις 14 Ιουνίου η Επιτροπή έκανε μία πρόταση και σχέδιο δράσης με 24 συστάσεις συγκεκριμένες για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος. Το σύστημα έγνος και η ανάπτυξή του αποτελούν σημαντικό μέρος αυτού του σχεδίου δράσης και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση. Θα πρέπει να τονίσουμε στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών ότι υπάρχει μέρος της αγοράς το οποίο καλύπτεται από τα ευφυή e συστήματα μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε κίνηση το σύστημα EGNUS ώστε να μπορεί να μεταδίδει εγγυημένα σήματα για την πολιτική αεροπορία και για να είναι σε αυτή τη στρατηγική σημασία αγορά ανταγωνιστική σε όλα τα επίπεδα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα EGNOS είναι συμβατό με το σύστημα GPS και θα προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες από το 2013 και μετά όταν θα τεθεί σε εφαρμοστή πλήρως τον Γαλιλαίο και είναι ανώτερο από το σύστημα GPS συνεργασία μεταξύ Galileo και GPS θα είναι θετική δεδομένου ότι θα υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων και θα βελτιωθεί η λειτουργία της. Το, το σχέδιο δράσης της Κομισιόν της 14ης Ιουνίου προβλέπει τις διάφορες τομεακές δράσεις και ξέρουμε ότι θα βοηθήσει ε, και για την ε, ολοκλήρωση της ενιαίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού θα βοηθήσει επίσης το σύστημα και την, ε, τον ναυτιλιακό τομέα, θα βοηθήσει τα οδικά συστήματα, την ε, διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων ε, για την ασφάλεια, για τους ταχογράφους, τους ηλεκτρονικούς, για τα συστήματα διοδίων και χάρη στα δεδομένα τα οποία θα περιέχει το GNSS θα γίνεται και καλύτερη, ε, θα υπάρχει καλύτερη εγγύηση και επαλήθευση των στοιχείων. Στην έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνονται σε σχέση με το Γαλιλαίο οι πρόεδροι που έχουν επιτευχθεί προβλέπεται η συνεργασία με τα άλλα συστήματα τα δορυφορικά και το σύστημα αυτό θα μπορέσει το GNSS και το Galileo να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο είναι και από οικονομικής πλευράς και από άποψη ασφάλεια των πολιτών πάρα πολύ σημαντικό για μας. Τώρα, τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Στην έκθεσή μας συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία στις δράσεις που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται θα πρέπει να γίνουν με συντονισμένο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις με ό,τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρουμε επίσης ότι δυστυχώς τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεπαρκή. Και αν θέλουμε να υποφεληθούμε από τα συστήματα έγκνος και Γαλιλαίο πλήρω, θα πρέπει να δημιουργήσουμε από τώρα υπηρεσίες και εφαρμογές που να σχετίζονται με τα συστήματα αυτά, ώστε όταν θα μπορέσουμε να τα θέσουμε σε λειτουργία, να υποφεληθούμε πλήρως από τις εφαρμογές αυτές. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να χορηγήσουν λοιπόν, να προβλέψουν τη χορήγηση των απαραίτητων κονδυλίων στα πλαίσια των, ε, μελλοντικών δημοσιονομικών οπτικών και στα πλαίσια των ετησίων προπολογισμών, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα στρατηγικής ε, σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρσι κάναμε στις αρχές Δεκεμβρίου μία μίνι ακρόαση Uh, Και καταλήξαμε σε δύο σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, μεταξύ των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπάρχει γενικότερο πρόβλημα κονδυλίων. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφτούν περισσότερα κονδύλια. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε όλα αυτά τα οποία προτείνουμε να γίνουν ελκυστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα μεταξύ όλων ότι θα υπάρχουν και κοινοτικά κονδύλια που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις αυτές. Υπάρχουν νέες διατάξεις που προβλέπονται για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική στα πλαίσια της νέας συνθήκης της Λισαβόνας. Και το Galileo και το GNNS, όπως είπα και επαναλαμβάνω, είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου η σημερινή έκθεση, πιστεύω ότι αποτελεί θέμα στρατηγικής σημασία σημαντικό για την τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την έκθεσή μου όλοι οι συνάδελφοι, ώστε να ζητήσουμε με σαφήνεια από την Επιτροπή μας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, και από το Συμβούλιο να υποστηρίξουν το σύστημα αυτό στα πλαίσια της... Σας ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ κυρία Τσικάου. Εκ μέρους του ΕΛΚ ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ την συνάδελφο για την έκθεση αυτή. Äh, Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι για μας ε, ότι εμείς ε, το ΕΛΚ συμφωνούμε με την έκθεση αυτή για το GNSS και τον Γαλιλαίο. Ε, οι διεκδικήσεις αν θέλετε απέναντι στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν είναι δικαιολογημένες δεν ε, έχουμε λόγο να περιμένουμε ε, μέχρι ότου να γίνουν ορισμένα πράγματα για να έχουμε τέλο πάντων κάποια επιστροφή από την ε, ε, από την επένδυση αυτή δεν νομίζω ότι είναι ε, λογικό αυτό έτσι και αλλιώς ε, περιμέναμε πολύ καιρό για τον Καλλιλέο εντωμεταξύ έχουμε 8 δις τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη και όσον αφορά τώρα το GNSS πραγματικά πιστεύουμε ότι ότι ε, θα προχωρήσουν τα συστήματα αυτά θα προχωρήσει το σύστημα ήδη έχουμε 24 ε, εκατομμύρια σε μερικά χρόνια θα έχουν διπλασιαστεί τα ποσά αυτά και οι ε, Αμερικανοί βεβαίως δουλεύουν ήδη, έχουν ε, υιοθετήσει το ε, GPS και τα λοιπά. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα ε, για τον ανταγωνισμό, να δημιουργηθεί αν θέλετε φοβερή την παράθεση ε, σε επίπεδο ανταγωνισμού. Ερώτηση προς την Κομισιόν βεβαίως τι γίνεται, τι κάνουν οι Κινέζοι. Τώρα, παρακάτω, η κυρία Τικάου λέει πάρα πολύ σωστά ότι στον τομέα των μεταφορών έχουμε συστήματα που υπάρχουν όμως διαφορετικά ε, Στι μεταφορέ γενικώ υπάρχουν πολλά συστήματα τα οποία προσπαθούμε όμως να τα γεφυρώσουμε. Εν τω μεταξύ όλα τα έσοδα που γίνονται στα διάφορα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξαναμπούν σε επενδύσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών ε, αυτό είναι το περίφημο earmarking που λέμε από εκεί και πέρα για τις θεσά, θαλάσσιες μεταφορές πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των σκαφών πώς μπορούμε σε ορισμένες θαλάσσιες διαδρομές θαλάσσιες οδούς όπως παραδείγματο χάρη στο Βόσπορο πώς μπορούμε να έχουμε ε, ακριβή συστήματα που να ελέγχουν τα πράγματα και τον Γαλιλαίο προσφέρει ένα τέτοιο επακριβές σύστημα για τις εναέρειες μεταφορές βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσουν περαιτέρω οι διαπραγματεύσεις με την ΙΚΑΟ για να έχουμε ε, σαφή εικόνα και εδώ τώρα ένα παράδειγμα εφαρμογής που το ζήτησαν και άλλοι τέσσερις ευρωβουλευτές είναι η εξέταση, επιθεώρηση αν θέλετε των ενισχύσεων και στις και γεωργικές δαπάνες γίνεται ε, αυτό και το ίδιο μπορεί να γίνει και εδώ όπως μετράμε εκτάσεις στη γεωργία μπορούμε και εδώ με αυτό το ακριβές σύστημα να έχουμε περισσότερη ασφάλεια και περισσότερη διαφάνεια Ευχα... κλείνοντας να ευχαριστήσω την κυρία Τικάου για την δουλειά που έκανε για την εξαιρετική αυτή έκθεση Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Άλντι, κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Τικάου. Νομίζω και εγώ ότι έκανε μια πολύ καλή έκθεση. Ε, ίσονος σημασίες παρατηρήσεις έχουμε. Όταν ε, φτιάχναμε το, το πρόγραμμα δράσης ITS για τις χερσές οδικές μεταφορές είχαμε πει ότι χρειάζεται προδιαγραφές για τις εφαρμογές του, του GNSS. Ε, αυτό βέβαια δεν προδίκαζε ότι οι εφαρμογές, αυτές ήταν εφαρμογές Γαλιλαίου. Αν είναι οι καλύτερες οι εφαρμογές Γαλιλαίου, εντάξει. Αλλά Όντως όπως ελέγχθη πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποιοι ήδη έχουν επενδύσει, άλλοι θέλουν να τραβήξουν το δικό τους δρόμο, αλλά εάν και εφόσον είναι όντως καλύτερες οι εφαρμογές καλλιλέω ας τις υποστηρίξουμε, θέλουμε όμως να εξασφαλίσουμε ότι είναι οι καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές. Εδώ λέγεται ότι οι Αμερικανοί ξοδεύουν 200 με 500 εκατομμύρια το χρόνο για εφαρμογές ενώ εμείς δαπανούμε 50 το 1 δέκατο είναι τεράστια η διαφορά και ε, Βεβαίω στην ανακοίνωση αναφερόταν και στην ανακοίνωση της Κομισιόν αναφερόταν και η ανάγκη να ε, βρεθούν επιπλέον κονδύλια. Αυτό είναι η δουλειά βέβαια της Επιτροπής Προϋπολογισμών να υπάρξει μια κάποια ελαστικότητα για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε κάποια κονδύλια εδώ. Ο κύριος Κούν είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν ορισμένα πράγματα στις θαλάσσιες μεταφορές και σε αέριες μεταφορές. Συμφωνώ, αλλά και στις οδικές μεταφορές θα ήθελα να τονίσω. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εδώ. Και υπάρχει και το θέμα της οδήγης και των ορών ανάπαυσης των οδηγών. Στη χώρα μου οι φορτεγατζίδες έχουν μάθει να πειράζουν αν θέλετε τους ταχυγράφους ε, οπότε γίνονται μεγάλες κομπίνες εκεί και συνεχώς προσπαθούμε να βρούμε καλύτερα συστήματα πιο πιο αξιόπιστα, δηλαδή που να μπορούν να ελέγχουν τι συμβαίνει για λόγους ασφάλειας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε, να υπάρχουν εφαρμογές του καλλιλέου να χρησιμοποιηθεί το καλλιλέο σαν εργαλείο για την α, ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οδικών μεταφορών, αλλά για να εξασφαλιστεί και καλύτερη ανάπαυση και λιγότερο στρες για αυτούς τους οδηγού των φορτηγών που εξυπηρετούν ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλο πάντων, για να μην μακρηγορώ, είμαι υπέρ τη προσέγγιση σα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο παραπάνω το θέμα των κονδυλίων τη χρηματοδότηση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό που η Κομισιόν ε, πρότεινε αυτό το σχέδιο δράση. Το χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ για τους πράσινους κυρία Λίχτενμπέρκερ. Ευχαριστώ πολύ. Για... Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Νομίζω ότι ελέγχθησαν πολλά πράγματα που δεν θέλω να επαναλάβω. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι η πτυχή της διαλειτουργικότητας. Αν αρχίσουμε να αγνοούμε την διαλειτουργικότητα ακόμη και αν αυτό δεν υποστηρίζει μονοπόλια αλλά ε, αγνοεί όμως ορισμένα, ορισμένες πτυχές και υποχρεώνει κάποιους να αγοράσουν καινούργια μηχανήματα αν την αγνοούμε λοιπόν εμείς τη διαλειτουργικότητα φαντάζεστε τι γίνεται αλλού γι' αυτό επειδή αυτό εγώ θεωρώ ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας είναι, βασικό σφάλμα για το οποίο ορισμένα πράγματα πήγαν στραβά στην Ευρώπη, γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ή έγιναν λάθη σε συνδυασμό και με την, ε, τις υποδομές και τα λοιπά. Ενώ οι Αμερικάνοι δεν έκαναν το λάθος αυτό και ήταν πολύ πιο αποτελεσματικοί. Όταν λέει η συνάδελφος Γιάννησεν ότι ορισμένοι ορισμένες χώρες ε, ε, χρηματοδοτούν και ε, δίνουν περισσότερα κονδύλια για άλλους, άλλες μεθόδους βέβαια για το GPS έχει δίκιο απ' την άλλη μεριά όμως ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη μεριά όμως τον Καλιλαίο έχει μια τεράστια πολιτική διάσταση. Και θα πρέπει να γνωρούμε βεβαίω και την, ε, το μεγάλο ποσοστό των στρατιωτικών εφαρμογών στις Ηνωμένε Πολιτείε που εμείς ούτε το έχουμε ούτε το θέλουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η, δια, η προτίμηση η επιλογή μεταξύ Γαλιλαίου και GPS καθίσταται πραγματικά τελείως πολιτική επιλογή και θα πρέπει να δούμε και τι θα κάνει και η Κίνα βεβαίως αλλά αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε την πολιτική διάσταση πρέπει να την έχουμε κατά νου και θα πρέπει να προσπαθήσουμε στην Ευρώπη να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ούτω ώστε οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται να είναι και ε, ε, πρακτικά και πραγματικά σωστές Αυτά γενικώ. Τώρα για τις κάποιες λεπτομέρειες, ιδιαίτερα για τις εφαρμογέ, εφαρμογές, θα πρέπει να προσέξουμε ε, στις οδικές εφαρμογές ε, ειδικά να προωθήσουμε και την ε, της ε, της ε, πολλαπλές ε, τις μεταφορές διαφόρων ειδών, τις συνδυασμένες μεταφορές. Για, γιατί αν ε, αυτό, μπορεί να μην βοηθάει ορισμένα μονοπόλια αλλά εμείς δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε τα μονοπόλια των χωρών μας και όπως είπα και πριν να δούμε λιγάκι παραπάνω το πτυχή χρηματοδότησης η Ευρώπη υστερεί εδώ γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε λίγο παραπάνω στην έκθεση το κομμάτι των κονδυλίων Ευχαριστώ πολύ κυρία Φώστερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Νομίζω θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυρία Τίκαου, διότι έκανε εξαιρετική δουλειά σε ένα τόσο περίπλοκο θέματα. Και είναι περίπλοκο και χρονοβόρο, διότι το έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση δεν έλαβε η χώρα την τελευταία φορά που είχαμε ζητήσει το θέμα αυτό και τώρα γίνεται. Αλλά υπάρχουν ακόμα διάφορα θέματα, διάφορες εκκρεμότητες. Αν δούμε όλα αυτά τα χρόνια που υποστηρίζαμε την εισαγωγή του Γαλιλαίου, του προγράμματος Γαλιλαίου, και δεν χρειάζεται να μπω σε όλους τους τομείς ε, που έχουν ε, καλυφθεί ε, και από άλλους ομιλητές, δηλαδή να μιλήσω για τα πλέον εκτήματα και τους τομείς που θα θίξει, αν θέλετε, που θα επηρεαστούν από το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης. Ε, αυτό το οποίο όμως παραμένει λίγο ασαφές για, για μένα και θα ήθελα κάποιες ε, πληροφορίες από την Κομισιό είναι τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Διότι αν ε, δούμε το, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, δεν ξέρουμε τι γίνεται και υπάρχει και μεγάλη έρευνα από τον ιδιωτικό τομέα. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε τέτοιου είδους project, τέτοιου μεγέθους, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, συνέχεια. Βέβαια υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία είναι πιο διαθέσιμα και πιο πρόθυμα από άλλα. Αλλά εάν είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει και τα κάνει σωστά τα πράγματα, είτε όχι. Διότι οι επενδύσεις, ε, όταν μιλάμε για έρευνα και ανάπτυξη, ε, όπως ε, πολύ σωστά ελέγχθη, είναι ε, μια διαδικασία ιδιαίτερα περίπλοκη, τουλάχιστον πιο περίπλοκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς δεν είμαστε στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα όμως τα πράγματα προχωρούν, δεν προχωρούμε, δεν προχωρούν, έρπουν αν θέλετε. και αυτό είναι ένα από τα μπουσουλάνε. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε για τα θέματα της χρηματοδότησης. Η Κομισιόν δεν ήταν σαφής. Γι' αυτό διαρωτώμε μήπω έχει να μα δώσει κάποιε περισσότερε λεπτομέρειε για το πώ θα προχωρήσουμε. Διότι χωρί αυτό δεν προχωρούμε. Φαίνεται ότι χρονοτριβούμε με συζητήσεις, συζητάμε που βρισκόμαστε, τι θα κάνουμε, αλλά το πρόβλημα είναι πού θα πάμε. Αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ο κύριος Κόλιτσεκ. Θα πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που η Επιτροπή μας προχωράει γρήγορα στις ε, συζητήσεις μας. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την συνεδρίαση από την αρχή και την ψηφοφορία της ε, έκθεσής μου την παρακολούθησα από το, αυτοκίνητό μου, διότι κόλλησα στην κυκλοφορία των Βρυξελών. Συμβαίνει, συμβαίνει αυτό στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, Ας επανέλθουμε στην έκθεσή μας. Να ευχαριστήσω την κυρία Τικάου για την τόσο καλή έκθεση εξαιρετικής ποιότητας. Ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν ε, στο κείμενο αυτό. Εμείς ε, ε, θέλουμε να εφαρμοστεί το σύστημα και θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους της Κομισιόν το εξής. Είναι αλήθεια ότι οι χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας ενδιαφέρονται για το project αυτό. Από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι ξέρω, οι ΙΔΙ ενδιαφερόντουσαν ιδιαίτερα πριν από κάνα δύο χρόνια. Επομένως θα μπορούσε η Κομισιό να επιτρέψει ε, κάπως στον Γαλιλαίο να συμμετέχει στα συστήματα πληροφορικής, ε, να μπορεί να εφαρμόζεται δηλαδή με τον καλύτερο, με το πιο εύκολο δυνατό τρόπο, να είναι φιλικό στο χρήστη. Ε, όλοι χρησιμοποιούμε λίγο πολύ τα περίπου ίδια κινητά, αλλά όλοι έχουν διαφορετικά ανταλλακτικά και προσπαθούμε να εναρμονίσουμε αυτό τον τομέα. Μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και εδώ μια τέτοια προσπάθεια, δηλαδή να ξεκινήσει το σύστημα με, με πιο ε, λογικό, αν θέλετε, τρόπο, πιο φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Και ο Γαλιλαίος να είναι, να είναι καλύτερος σε αυτόν τον τομέα από ό,τι τα ανταγωνιστικά συστήματα. Υπάρχει μία προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στην Κόνας και στο Γαλιλαίο θα, στο GNSS δηλαδή και στο Γαλιλαίο. Και Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι εισηγητέ. Μιλάω για συμβατότητα ανάμεσα στο έγνος και στο Γαλιλαίο κυρίως, Κατά τα λοιπά, συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες ε, και θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ καλά και περιμένουμε με ενδιαφέρον την συνέχεια όλου αυτού του project. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τικάο για την εξαιρετική ποιότητα της εκθεσής της και θα ήθελα να πω κάτι για ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση και το έθιξε και η κυρία Γιάντσιν η διαφορά ανάμεσα στον Γαλιλαίο, στο GPS ή στο Κινέζικο είναι ότι εδώ μιλάμε για ε, πολιτική χρήση αν θέλετε, ενώ τα άλλα είναι για στρατιωτική χρήση. Και δίνουμε συνήθως πάρα πολλά χρήματα για να στείλουμε ε, χρήματα στο στρατιωτικό τομέα, αλλά πολύ λιγότερα χρήματα για να ε, μπορούν να κινηθούν τα πλοία μας ε, ή τα αεροπλάνα μας σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει και ένα θέμα μορατόριου, αν θέλετε, διότι προχωράμε, βρίσκουμε τα χρήματα ε, και προχωράμε. Αν δεν τα βρούμε, τι γίνεται, σταματάμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ρυθμίσουμε. Επίση, ε, είναι και ένα άλλο σημείο το οποίο με ανησυχεί και θα πρέπει να ρυθμιστεί και την έκθεση και να μα απαντήσει η Κομισιό, το κόστο λειτουργία. Από τη στιγμή που εφαρμοστεί το, το σύστημα, κοστίζει, διότι πρέπει να το συντηρούμε, θα πρέπει να το ανακαινίζουμε και θα υπάρχουν ε, θα υπάρχει κόστος. Εάν αυτό το κόστος είναι αρκετά χρήματα, εκατοντάδες ή εκατομμύρια ευρώ ε, κάθε χρόνο, μήπως θα πρέπει να ενδιαφερθούμε για το πόσο χρηματοδοτηθεί αυτό το κόστος. Δηλαδή, είτε η Κομισιόν και οι αρμόδιες ε, επιτροπές, η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα φροντίσει έτσι ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του Γαλιλαίου, το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερα καινοτόμο για το, σύστημα, το δημοσιονομικό μας σύστημα, ή θα προβλέψουμε ότι υπάρχουν έσοδα γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε θίξει. Έσοδα από την ε, εκμετάλλευση, πολιτική εκμετάλλευση του Γαλιλαίου. Και από τα έσοδα αυτά θα χρηματοδοτηθεί η συντήρηση και η ανακαίνιση του Γαλιλαίου. Και εδώ τίθεται θέμα ιδίων πόρων της Ευρώπης, που είναι μια άλλη δημοσιονομική συζήτηση στην Ευρώπη και, και ε, απευθύνομαι στην κυρία Γένσεν. Γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, ήδη, αν μπορώ να το πω, Ξεκινήσαμε με ένα προπολογισμό ο οποίος θα τριπλασιαστεί από ό,τι φαίνεται μέχρι και συνεχίζουμε να μην μιλάμε για τη χρηματοδότηση, ενώ οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και για την συνέχεια της ζωής του Γκολιλαίου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο να ε, προβλέπουμε να ρυθμιστούν τα θέματα προπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι τι θα γίνει, πολύ σημαντικό αυτό, τι θα γίνει με τον Γαλιλαίο ε, όσον αφορά τη συντήρηση και την αγκέννηση του μετά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόσκο από την Κομισιό έχει το λόγο. Καλημέρα σας κύριε Συγήτρια, κύριε Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι μέλη της Επιτροπής σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Τσικάου για το σχέδιο έκθεσης, το οποίο είναι εξαιρετικό και αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των εφαρμογών του GNSS. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το γεγονό ότι τονίζει πόσο σημαντικά είναι τα συστήματα αυτά υπάρχει τη γεωστατική πλοήγηση. Γνωρίζουμε ότι στις ε, μεταφορές ε, αυτά τα συστήματα πλοήγησης είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον. Είμαστε βεβαίως ε, υπέρ του σχεδίου δράσης, το οποίο παρουσιάσαμε και όπως περιγράφεται και στο σχέδιο δράσης θέλουμε η τομεακές δράσεις να ε, εφαρμοστούν ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα για την δορυφορική ραδιοπλοήγηση. Για να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν, θα πω πρώτα απ' όλα ότι όταν αναφορά την ε, υποδομή και την εφαρμογή του συστήματος, συνεχίζουμε τις εργασίες μας παρούσα χρηματοδότηση στα πλαίσια των προϋπολογισμού σήμερα μας επιτρέπουν να ολοκληρώσουμε έως το τέλος της παρούσας διαδικασίας προϋπολογισμού την οργάνωση 18 ε, τέτοιων έργων υποδομής. Η, το θέμα της ε, λειτουργίας περαιτέρω θα συζητηθεί στα πλαίσια της προσωρινής μέσω πρόθεσμης ε, αναθεώρησης. Θα πρέπει να μελετήσει το όλο θέμα η Επιτροπή και να απαντήσει. Για να απαντήσω συγκεκριμένα τώρα σε ένα θέμα που τέθηκε, ο προϋπολογισμός λειτουργίας, έτσι όπως προβλέπεται, ε, στα πλαίσια της προσωρινής αναθεώρηση είναι 800 εκατομμύρια ευρώ ετηρίως. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας για να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω η υποδομή με την ε, Ευρωπαϊκή Εθνική Υπηρεσία, αλλά και με τους συνεργάτες μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις ε, συχνότητες συνεχίζονται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη ή διμερός ή πολυμερός με τρόπο ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες και εδώ αναφέρομαι κυρίως τους Κινέζους αλλά και στους Ρώσους, τους Ιάπωνες, τους Ινδούς και αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι γίνονται και τεχνικού επίπεδου συζητήσεις και με τους συναδέλφους τους Ινδούς για τις συχνότητες αλλά και βεβαίως με τους Αμερικανούς, τις GPS με τους οποίους έχουμε υπερβεί το στάδιο των συζητήσεων για την συμβατότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά σε κάθε σύστημα, ώστε να μην υπάρχουν παρεμβάσει με άλλα συστήματα. Το ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο, είναι και εκτιμένο, αλλά συζητούμε με τους Αμερικανούς και για διαλειτουργικότητα, δηλαδή για την δυνατότητα τα δύο συστήματα να εποφελούνται αμοιβαίω. Δηλαδή οι δορυφόροι του ενός θα μπορούσαν να τροφοδοτούν με στοιχεία ή να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση στοιχείων του άλλου. Νομίζω ότι έτσι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις που αφορούν τις υποδομές. Εάν ε, δεν ε, ήμουν αρκετά ακριβής μπορώ να επανέλθω τώρα για να φτάσω στην έκθεση και στο θέμα των εφαρμογών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πούμε στην έκθεση της κυρίας Τσικάου ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη. Οι εφαρμογές GNSS είναι ένας τομέας στον οποίο παρατηρείται όντως ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή εκ μέρους των ΜΜΕ σε σχέση με άλλους τομείς και ένα μέρος της χρηματοδότησης πρέπει να δω ότι είναι μάλλον η αναλογία της χρηματοδότησης εδώ είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με άλλους τομείς. Έχουμε λοιπόν έλλειμμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως αναφέρει και η έκθεση, θα πρέπει να διορθώσουμε να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση και συμφωνούμε βεβαίως με αυτή την άποψη. Επίσης, ε, μία από τις δράσεις, μία τις δράσεις του σχεδίου δράσης αναφέρει τις προσπάθειες που έχουν αρχίσει και εκ μέρους της Κομισιόν ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν συνεργασίες, συνεργείς για να γίνουν κάποια πράγματα από κοινού κυρίως σε θέματα εφαρμογών στην θέμα των τεχνολογιών και των GMS όπως αναφέρεται. Αναμένουμε λοιπόν την τελική εκδοχή της έκθεσης της κυρίας Τσικάου που πιστεύουμε ότι είναι μια σημαντική υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό, κυρίως για την ε, ε, ανάπτυξη του συστήματος ΑΒΑΛ που βασίζεται στην ε, ανάπτυξη του ε, συστήματος GPS. Η κυρία Τσικάου, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν το λόγο. Θα περιμένω τις τροπολογίες που θα θελήσουν να καταθέσουν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να παραλαμβάνω πόσο μεγάλη στρατηγική σημασία είναι για την Ευρώπη η ανάπτυξη του συστήματος έγνος και γαλιλαίο όσον αφορά την χρηματοδότηση. Επιτούτης, σε αυτή την αρχική έκθεσή μου δεν ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένη, διότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί πρώτα απ' όλα η προσωρινή μεσοπρόθενη αναθεώρηση και περιμένουμε στα πλαίσια των προσεχών δημοσιονομικών προπτικών να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις τις οποίες θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσα να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δεν επέμεινα τώρα. Σίγουρα θα υπάρξουν τροπολογίες σε σχέση, εκ μέσω συναδέλφων σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Και... Βεβαίως θα θέλαμε να υπάρξει, ε, και αυτό θα αποτελέσει θέμα των τροπολογιών, πρόταση για να αυξηθεί η χρηματοδότηση που προβλέπετε εδώ. Στην ε, έκθεση μου αυτή, όπως σας είπα, δεν ε, ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένη διότι ελπίζω ότι θα υπάρξουν σχετικές πρωτοτροπολογίες. Το σύστημα Γκαλιλαίο για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, κυρίως όσον αφορά τις αδετικές μεταφορές, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα σύστημα ε, τεχνολογίας. Θέλουμε να υπάρξει συνεργασία. Γι' αυτό περιμένουμε προτάσεις και εξελίξεις και περιμένουμε να ολοκληρωθούν και τα διάφορα έργα υποδομής. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπαμε, το σύστημα έγνωσης θα πρέπει να μπορέσει να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μπορέσει να εφαρμοστεί το σύστημα έγνωσης και βόρεια και δυτικά και νοτιο Αυτή τη στιγμή η κάλυψη σε αυτές τις περιοχές δεν είναι επαρκής. Μιλούμε για ενιαία αγορά και πιστεύω ότι είναι στρατηγική σημασίας ο Βορράς, ο Νότος και η Ανατολική πλευρά της Ευρώπης να καλύπτονται καλύτερα. Γι' αυτό θα ήθελα κυρίως να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρητά να λάβει υπόψη αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Τσικάου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 8 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε την της κυρίας Τσικάου το Μάρτιο και στην Ολομέλεια του Μαΐου. Οκτώ λοιπόν είναι και πάλι ε, Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνω μία κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα της επιμερήσης διάταξης επιβολή τελών στα, βαρέα, στα βαρέα φορτηγά του κυρίου Ελ Καντράουι. Κύριε Καντράουι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Περιμέναμε δύο χρόνια τη θέση του Συμβουλίου Τώρα πια έφτασε η στιγμή λοιπόν να κάνουμε ένα κάποιο βήμα προς τα μπρος διότι όπως θα ξέρετε το Συμβούλιο πήρε απόφαση και έτσι θα πάμε στη δεύτερη ανάγνωση κι εμείς. Τώρα πριν να μπω σε λεπτομέρειες να σας πω μερικά πράγματα για τις δυσκολίες των διαπραγματεύσεων. Στην αρχή το Συμβούλιο υιοθέτησε μία κοινή θέση αλλά με ελάχιστη πλειοψηφία ρω τρεις ψήφοι ήταν η διαφορά ε, Πρώτη δυσκολία λοιπόν αυτή, δεύτερη, κατά την πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα κείμενο το οποίο ήταν πολύ πιο φιλόδοξο από το αρχικό κείμενο αλλά και πάλι η πλειοψηφία ήταν πολύ μικρή. Αυτό όλα σημαίνουν αγαπητοί συνάδελφοι ότι αν θέλουμε τα πράγματα να γίνουν πιο φιλόδοξα από ό,τι ήταν αρχικά θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία για την ε, ε, για ε, για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε την άποψη αυτή. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να πολλές πολιτικές ομάδες να υποστηρίξουν ε, μια φιλόδοξη θέση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα το ερώτημα θέλουμε συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση ή θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία κατά την οποία θα περάσουμε ό,τι μπορούμε στη δεύτερη αναγνώση αλλά <coughs> θα μπούμε στη δύσκολη διαπραγμα... ε, διαδικασία της συμφιλίωσης Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι υπάρχουν προθεσμίες τις οποίες πρέπει να τηρήσει το Κοινοβούλιο και βεβαίως το θα πρέπει να ε, θα, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε 16 Φεβρουαρίου πάει το κείμενο στην Ολομέλεια αν έχουμε τέσσερι μήνες μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να βιαστούμε <coughs> αλλά ήδη μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν προχωρήσει πολλά πράγματα όπως καταλαβαίνετε τροπολογίες, ψηφοφορίες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, οι, διαδικασία είναι, οι διαδικασίες είναι δύσκολες. Και τώρα για να δούμε το περιεχόμενο της έκθεσης. Το Συμβούλιο έχει όπως σας είπα πάρει κάποια θέση αλλά ε, με την οποία εμείς διαφωνούμε. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Ε, ε, η αρχή βέβαια της λήψη υπόψη των του εξωτερικού κόστους και ένταξη του εξωτερικού κόστους σε κάποια πράγματα αυτή η αρχή έχει γίνει αποδεκτή αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες στις οποίες διαφωνούμε. Η, το, το θέμα είναι τι ορίζουμε σαν εξωτερικό κόστος, γιατί η Κομισιόν δίνει διαφορετικό ορισμό από ό,τι εμείς. Το Συμβούλιο έχει μελετήσει, επίσης, έχει μελετήσει τις υποδομές και θέλει να αλλάξει ορισμένα πράγματα ε, στις υποδομές σε σχέση με αυτά που υποστηρίζουμε εμείς και η Κομισιόν. Εμείς λέμε ότι η ένταξη η μετατροπή αν θέλετε των εξωτερικών δαπανών σε εσωτερικές δαπάνες δεν θα πρέπει να είναι ένα είδος φορολογίας ε, η θέση του Συμβουλίου είναι διαφορετική. Το Συμβούλιο βεβαίως ε, αυτού απλώς θα κάνει μια ε, θα, θα είναι αρκετά ευέλικτο και θα ζητήσει να είναι προερωτικά αυτά εμείς θέλουμε να γίνουν προϋποχρεωτικά μιλάμε για οδηγία έτσι κι αλλιώς Πολλά βεβαίω από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν εμάς δεν τα έχει λάβει υπόψη η Κομισιόν ή παίζει ρόλο η διαλειτουργικότητα δεν λαμβάνεται υπόψη εδώ απαρκώς τα, ο υπολογισμό του κόστους ανά χιλιόμετρο κτλ. Και ε, εδώ ε, θα πρέπει να ε, βρούμε τρόπους να προσεγγίσουμε οι μεν τους δε. Έχω κάποιες προτάσεις εγώ προσωπικά που θα ήθελα να τις παρουσιάσω για να δω τι πιστεύετε κι εσείς. Πρώτα-πρώτα έχουμε ε, κάποια θέματα όπως παραδείγματο χάρη το τέλος συμφόρησης το congestion charge το οποίο διαφωνούμε με τη θέση του Συμβουλίου εδώ δεν είναι σίγουρα δύσκολα θα συμφωνήσουμε. Φοβάμαι. Ε, κάποιες πολιτικές ομάδες βεβαίως θέλουν να συνδυάσουν, να συνδέσουν το τέλος αυτό με τα γιοταχή. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει αυτό. Θα πρέπει να δούμε ε, τι γενικότερο το θέμα των τελών υποδομής και πώς μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα εκεί. Οι δυνατότητες που έχουμε δεν είναι και πάρα πολλές. Ε, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το τέλος αυτό το Συμβούλιο ζητεί αύξηση κατά 175% αυτού του είδους των τελών ε, μιλάει για πέντε μέρες, πέντε ώρες την ημέρα το Συμβούλιο σαν οριακό χρόνο αλλά δεν ξέρω εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε αν θέλετε το τέλος συμφόρησης με άλλα θέματα στα οποία μπορεί να ζητήσουμε παραπάνω ευελιξία. Εμά eh, principe moet aanvaard worden, zodanig dat... μας ενδιαφέρει εδώ να βοηθηθεί και ο καταναλωτής των φορτηγών, αν θέλετε, τον, ε, όχι μόνο ο οδηγός του Ιωταχή υπάρχουν τέλος πάντων διαφορετικές απόψεις αλλά για, αυτό το, για αυτή την πρώτη δέσμη μέτρων νομίζω ότι πρέπει να επιζητήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Βεβαίως θα χρειαστεί αναθεώρηση των μέτρων αυτών σε μερικά χρόνια, αυτό το έχουμε υπόψη μας. Τώρα, προχωρούμε στο δεύτερο θέμα Τα θέματα της χρηματοδότησης τώρα. Θα τα συζητήσει αυτά το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι άσπρες ή μαύρες. Υπάρχουν πάρα πολλές διαβαθμίσεις του γκρι. Θα πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε ευελιξία, τη διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε συμφωνία ούτε καν στην ε, διαδικασία συμφιλίωσης. Ούτως ή άλλως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποδεχθεί να μην ευρεθεί λύση στο θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί να δούμε ποιο είναι το κεκτημένο και από νοθοτημοθετικής πλευράς, ποια είναι τα κονδύλια που προβλέπονται, τι γίνεται με τα θέματα ανταλλαγής και εμπορίας των, και τα δικαιώματα των εκπομπών. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουν όλα αυτά τα μέτρα να βοηθήσουν στη βελτίωση των συστημάτων. Θα πρέπει λοιπόν στην οδηγία για την ε, Ευρωβινιέτα να δεχθούμε ένα μέρος των εσόδων να συνηφέρουν στην μείωση του εξωτερικού κόστους. Επίσης να δούμε τι θα γίνει με τα διευρωπαϊκά προγράμματα και με τα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και νέα συστήματα χρηματοδότησης των υποδομών. Θα πρέπει επίσης να δούμε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των κρατών μελών. Διότι αν επιβάλλουν κάποια τέλη, θα πρέπει να μας πούν ποια είναι η χρήση τους. Για πού προορίζονται τα κονδύλια αυτά πριν να αρχίσει να εφαρμόζεται το κάθε σύστημα. Αυτό ώστε να ξέρουν κάθε φορά οι χρήστες πού πηγαίνουν τα χρήματά τους και αυτοί που χειρίζονται βεβαίως τα έργα υποδομής να γνωρίζουν συγκεκριμένα, συγκεκριμένα ποια κονδύλια έχουν. Αυτό είναι ένα δεύτερο πακέτο μέτρων. Αν θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις μπορώ να είμαι ακόμη πιο συγκεκριμένος. Τρίτος άξονας. Ο άξονας ο οποίος ε, αφορά τα διάφορα οχήματα. Ποια οχήματα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν κάποιο τέλος σε σχέση με το πόσο ρηπαίνουν. Εκτός από το εξωτερικό κόστος είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο συμπληρωματικό τέλος το οποίο να προβλέπετε για κάποιες ορεινές περιοχές και μία αύξηση ενδεχομένω των τελών όταν θα πρέπει να ε, χρηματοδοτηθούν κάποια, κάποια έργα εναλλακτικών υποδομών. Όσο περισσότερο μιλάτε, τόσο περισσότερο πολύπλοκα γίνονται τα πράγματα, λέει ο πρόεδρος. Κάπου πρέπει να τελειώσετε, γιατί μιλάτε εδώ και 25 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε λίγο χρόνο ακόμη. Τελειώνω, λέει ο εισηγητή. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιους ευρωπαϊκούς κανόνες, κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμοστούν και για τις οποίες έχει δοθεί συμπληρωματικός χρόνος για την καταβολή τελών εκ μέρους των φορτηγών, των βαρέων οχημάτων. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα ώστε να μπορέσει να ανανεωθεί και ο στόλος των οχημάτων αυτών. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε το 2018. Τώρα, όπως θα ε, θυμάστε ίσως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006 πέτυχε μια νέα οδηγία το 2008. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε διαστάσεις ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και εδώ για άλλους ε, τρόπους μεταφοράς μια νέα οδηγία και άλλους τρόπους ώστε να μπορέσουμε να εσωτερικεύσουμε κατά κάποιο τρόπο το κόστος. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Και αν μπορέσουμε να επιτύχουμε συνένεση. Θα ήθελα στις αρχές Φεβρουαρίου να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τριμερή διάλογο με την Κομισιό και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με το Συμβούλιο, συγγνώμη, ώστε να δούμε ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Σε ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε εκτενή κατάλογο συναδέλφων που θέλουν το λόγο, γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Σκιώδης 4 λεπτά, οι υπόλοιποι συνάδελφοι 2 λεπτά για να ακούσουμε και την Κομισιό και να μπορέσει ο κύριος Αλ Καντράουι στο τέλος να απαντήσει. Η κυρία τον για 4 λεπτά, είπα οι σκιώδεις εισηγητές 4 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θα απαντήσω στον Σαΐτ στη γλώσσα του. Ώστε να μπορούμε να συνεννοούμεθα απευθείας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τον ευχαριστήσω για τον πραγματισμό τον οποίο επιδεικνύει όταν αναφέρεται στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι συμφωνώ μαζί του με, αυτό που είπε. Δηλαδή το ότι γενικά, σε γενικές γραμμές δηλαδή, το Συμβούλιο φαίνεται να πηγαίνει προς την ε, σωστή κατεύθυνση παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημεία ακόμη κάπως ασαφή. Θα πρέπει ούτως ή άλλως να αποσαφηνίσει για πολλά σημεία τη θέση του Ευρωπαϊκού ε, το Συμβούλιο. Κυρίως για... Αυτό το οποίο αναφέρεται στο εξωτερικό κόστος. Επίσης, το θέμα των ωραρίων είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Επίσης, τι σημαίνει διαφοροποίηση της τιμής των διοδίων εκτός ορών ε, ε, συμφόρησης. Μπορεί να υπάρξει αύξηση έσως και μέχρι 300%. Θα πρέπει το μέτρο να μπορεί να είναι ελκυστικό ώστε να αποφεύγονται οι συμφορήσεις κυκλοφοριακές. Για Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για τους εθνικούς και για τους διεθνείς μεταφορείς. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά ώστε να μην υπάρχει και διαφοροποίηση σε επίπεδο αμοιβών των μεταφορέων αλλά θα πρέπει βεβαίως κάτι να κάνουμε ώστε να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Επίσης, τα έσοδα. Τα έσοδα θα πρέπει να μας πει από αυτά τα διόδια το κάθε κράτος, ο κάθε υπεύθυνο φορέας. Τι θα τα κάνει, πού θα πάνε. Θα ήθελα να προτείνω για το θέμα αυτό των ε, πόρων των συμπληρωματικών που θα συμπληρωμαθούν και το πού θα πάνε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, το θέμα της διαλειτουργικότητας είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το λύσουμε. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα διαλειτουργικότητας, θα πρέπει όλα τα προβλήματα να λυθούν, όλες οι δυσκολίες που έχουν να ξεπεραστούν Την πρότασή του λέει το Συμβούλιο ότι δεν θα πρέπει να έχουμε αυξήσεις επί αυξήσεων και θα ήθελα να έχω για το θέμα αυτό περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όντως να ενθαρρύνουμε όλες τις επιχειρήσεις να αγοράσουν πιο καθαρά οχήματα. Επίσης, είπατε ότι θα θέλετε να υπάρχει τριμερής διάλογος ανεπίσημος τον Φεβρουάριο. Ποια θα είναι η θέση σου. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε για την ε, θέση αυτή που θα διαμορφωθεί μεταξύ μας και να ξέρουμε ποια είναι τα σημεία τα οποία θα συζητήσεις. Θα υπάρχει λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει σαφής έντολη εκ μέρους μας. Ευχαριστώ κύριο Στέρξ. Ευχαριστώ τον Σαΐντα για τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις που έκανα. Επιτέλους έχουμε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση. Το βασικό είναι να ξέρουμε τι θέλουμε, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συμφωνία και το σημαντικό είναι να συμφωνήσουμε επί της αρχής. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα παράδειγμα και ένα πρότυπο και για τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο, κυρίως όσον αφορά τον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους. Είναι ουσιαστική σημασία. Υπάρχει αυτή η διακύμανση, αυτή η δυνατότητα Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η δυνατότητα τέλους επί της κυκλοφορίας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το επιβάλλουμε. Ε, θα πρέπει να μιλάμε για την ίδια διαδρομή. Ε, τα κράτη-μέλη τι κάνουν, τι ε, έχουν υιοθετήσει, τι ρυθμίσεις έχουν υιοθετήσει. Επίσης το πέρασμα από 5 έως 8 ώρες. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Υπάρχει επίσης και ένα ουδέτερο όριο το οποίο ορίζεται ή θα πρέπει να υπάρχει ε, μια, ένα συντονισμό ή θα πρέπει να κάνουμε μια, ένα, ένα, συμψηφισμό ανάμεσα στα διάφορα φορτία. Επίσης, για την διαφορά ανάμεσα στο εξωτερικό κόστος και την, τα κόστο, το κόστος υποδομός. Αυτό θα πρέπει να είναι ουδέτερο κανονικά, μηδενικό. Πρέπει να διευκρινιστούν τα πράγματα. Επίσης, όσον αφορά την διαλειτουργικότητα, η οποία έχει εξαφανιστεί σε σχέση με αυτό που λέει το Συμβούλιο, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να ε, πανέλθει στο κείμενο. Είναι απαράδεκτο το σημείο αυτό να παραμείνει σε, έτσι σε κρεμότητα. Τώρα για τις ε, εξαιρέσεις ε, ρο 5, 6, πρέπει να σας πω ότι δεν σημαίνει ότι υπάρχει το Euro 6 για τα οχήματα, για τα βαρέα οχήματα, ότι εθαρρύνουμε ε, κάποιες εταιρείες να αλλάξουν, κάποια κράτη να αλλάξουν ε, το πάρκο οχημάτων τους. ενθαρρύνουμε, δεν υποχρεώνουμε. Τώρα σε σχέση με αυτό που είπε η συνάδελφος Βόρτμαν Κόλ. Θα πρέπει μέσω των, των τροπολογιών να μπορούμε να επηρεάσουμε το Συμβούλιο. Διότι σε σχέση με την πρώτη ανάγνωση έχει αλλάξει η σύνθεση του ε, Κοινοβουλίου και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ και να θυμηθείτε τα τέσσερα λεπτά. Ναι, εμένα όμως μονάχα μου το λέτε, όχι στους άλλους. Αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι καταρχάς ευχαριστούμε τον Σαΐντι για την έκθεσή του. Αν δείτε την θέση του Συμβουλίου, πρέπει να σας πω ότι με πιάνει κατάθλιψη διότι αυτό το οποίο παραμένει είναι θέματα αρχής. Τίποτε άλλο όμως το οποίο να μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τις μεταφορές. Ε, αν οι συνάδελφοί μου από τις κάτω χώρες και το Βέλγιο μιλάνε για ουδετερότητα, δεν θέλουν να υπάρχει κανένα κόστος στο δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν θα αλλάξει. Είπε μίλησε, μίλησε για ουδετερότητα στο κόστος. Αυτό το οποίο θέλω να πω εδώ, συνεχίζει η κυρία Λίχτενμπέργκερ στα γερμανικά, είναι ότι εάν ε, θέλουμε να ακολουθήσουμε την θέση, να επηρεάσουμε τη θέση του Συμβουλίου, θα πρέπει να καταλήξουμε, θα μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Για τα επιμέρους θέματα τώρα, νομίζω ότι κάποια θέματα με το Συμβούλιο δεν μπορούμε να τα πετύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν, ε, ειδικά για τη συμφόρηση του χάρη, για τα τέλη συμφόρηση, δεν τα βγάζουμε πέρα και με το Συμβούλιο. ας πάει στη συμφιλίωση η συμφόρηση δεν ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα αυτό βέβαια Άλλοι πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικό Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονό ότι εδώ ακριβώς για τα, τη συμφόρηση μπορούμε κάτι τι να κερδίσουμε αλλά εκείνο το οποίο εμένα μου φαίνεται πολύ σημαντικό είναι οι δείκτες. Δηλαδή αν υπολογίσουμε τι σημαίνουν αυτά που λέγονται εδώ σε ορισμένες περιπτώσεις η επιβα... επιβάρυνση στο περιβάλλον άμα συμπεριλάβουμε και θόρυβο και τα λοιπά ε, ε, για τις περιπτώσεις συμφόρησης έτσι αυτά ε, η επιβάρυνση είναι πολύ μεγάλη και θα πρέπει να τονιστεί πολύ περισσότερο ε. για μένα λοιπόν οι δείκτες μάλλον οι πολλαπλασιαστές για κάποια στοιχεία ε, που αναφέρονται εδώ ε, είναι πολύ σημαντικοί και, δεν, και θα πρέπει να τονιστούν για να μην εξαφανιστούν πίσω από τις συζητήσεις για τα τέλη και το για πόση ώρα θα ισχύουν τα τέλη αυτά. Θα είναι υποχρεωτικά τα τέλη αυτά. Ε, στην, ε, να πω κάτι άλλο. Υπάρχει μια Υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις στο αρχικό κείμενο που μας υποβλήθηκε, αρκετά σολομόντιες θα έλεγα, που βοηθούν τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να αλλάξουν ε, τη χρηματοδότηση ή τα, τους προϋπολογισμούς τους για να αλλάξουν το σύστημα χρηματοδότησης ε, βοηθούν τα κράτη αυτά αμένα αλλά ίσως δεν αρκούν τέλος πάντων <coughs> νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τη χρηματοδότηση, τα δικαιώματα εκπομπών Εντάξει, θα καταλαβαίνω τα δικαιώματα εκπομπών, αλλά εμείς θέλουμε να βοηθηθούν οι πολίτες και οι πολίτες θα βοηθηθούν άμα οι, οι, υπάρξουν κάποιες υποδομές αν θέλετε ε, σκληρές Τώρα, εκείνο που είναι σημαντικό το θέμα είναι επίσης το θέμα των markups, ε, των ε, επιπλέον χρεώσεων, συμπληρωματικών χρεώσεων. Ε, θέλουμε συνολικά να έχουμε ουδέτερο αποτέλεσμα ε, και γι' αυτό εδώ πρέπει να προσέξουμε για τα markup. Και άλλο ένα θέμα που είναι σημαντικό είναι οι 3,5 τόνοι. Αυτά είναι για μένα σοβαρά θέματα. Το earmarking θα μπορούσαμε να το δώσουμε στο Συμβούλιο αν θέλετε και θα μπορούσαμε να, υπολογι... να υποχωρήσουμε αλλά όχι για τις 3,5 τόνους. Λοιπόν, επόμενος ο, ο μιλητής ο κύριος Ζήλη αλλά διατηρήστε το χρόνο θα συνεχίσουμε βέβαια τις προσπάθειες συντονισμού που ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος όσον αφορά ε, το συμβιβασμό με την συμβαστική λύση με το ε, Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι πέντε τα σημεία, δεν χρειάζεται να τα να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω νομίζω τα θίξαμε αυτά και στη συνάντηση που είχαμε, υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή πλειοψηφία στο Συμβούλιο που πιστεύει ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία. Και αν το εφαρμόσουμε αυτό σε νέα θέματα, τελικά δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε οτιδήποτε στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι πιο μετριοπαθήσει και θα εξηγήσω ποιους, σε ποιους τομείς πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση. Καταρχάς η δυνατότητα που υπάρχει εσωτερικοποίηση του εξωτερικού χρέους και που αφορά την ε, συμφόρηση, την κυκλοφοριακή συμφόρηση θα μπορούσαμε να έχουμε μια συζήτηση όσον αφορά τις ώρες εχμής. Είναι 5, είναι 6, 150%, 200%, ποια θα είναι τα όρια δηλαδή ε, ε, τα οποία θα πρέπει να, τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Αυτά είναι και δεν μπορούμε να τα περιορίσουμε. Τώρα το earmarking πιστεύω θα μπορούσαμε να είμαστε πιο δραστήρια αν θέλετε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι, Υπουργοί Οικονομικών των Κρατών Μελών θα έχουν το λόγο τους να πούνε, αλλά και εμείς όμως θα πρέπει να παραμείνουμε στις θέσεις μας. Όσον αφορά την τα ευρωπαϊκή ταξινόμηση, οι κλάσεις 5 και 6 είναι σωστές, υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη, ε, κυρίως όσον αφορά το φορτίο για τις περιφερειακές χώρες, ε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανανεωθεί το ε, πάρκο των φορτηγών τα επόμενα χρόνια. Ε, θα επηρεαστεί η αγορά και αυτό αφορά και το Aero 5 και το Aero 5 και το Aero 6. Τώρα, για τους 12 τόνους, ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Εάν τονίσουμε ότι οι 3,5, τόνοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στο μέλλον, δεν θα επιτρέψουμε στην περίπτωση αυτή, κατά την ταπεινή μου άποψη, στην αγορά, για τα οχήματα, αν τα οχήματα, τα φορτηγά ε, μέχρι 12 τόνους έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις θαλάσσιες μεταφορές ή την εσωτερική ναυσιπλοεία, τα ποτάμια δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τότε για τα, ε, για τα οχήματα των 3,5 τόνων και όχι των 12. Τώρα, για το κριτήριο χρόνου απόστασης. Συμφωνώ με το Συμβούλιο ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κριτήριο χρόνου, ε, ας πούμε στην, ε, στις χώρες της Βαλτικής. Είχαμε μια συνάντηση, αν έχουμε ένα... όχημα το οποίο κυκλοφορεί ε, και μολύνει και τον ε, ε, προκαλεί και έχει ρήπανση και ατμοσφαιρική ρήπανση δεν μπορούμε να το κάνουμε ευχαριστώ να μιλήσω λιγότερο από τέσσερα λεπτά μπορώ ή τέσσερα λεπτά πρέπει οπωσδήποτε τέλος πάντων πιστεύω λέει ο κύριος Κόλουτσεκ ότι οι συνάδελφοί μας έχουν απόλυτο δίκαιο όταν λένε ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα και θα πρέπει να υπολογίσουμε το ε, εξωτερικό κόστος ε, για τη συμφόρεση δεν ξέρω αν θα, είμαστε, αν θα πετύχουμε ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ας πούμε, το, τα, εθνικά, η εθνική δρυμή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πώς θα περνάνε οι δρόμοι και τα λοιπά, τα φορτηγά και δεν ξέρω τι άλλο. Ε, για τη διαλειτουργικότητα επίσης, γι' αυτό το είχα θίξει και, στο, και στον Καλλιλέο. Ε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί το σύστημα πλοήγησης και εδώ. Διαφωνώ όμως με τον προηγούμενο μιλητή, ο οποίος είπε ότι τα 5, 6 ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από όλους και να θίξουμε το όριο των 3,5 τόνων. Πιστεύω ότι είναι λογικό το όριο και θα πρέπει να επιμείνουμε. Επίσης θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα φορτηγά θα πρέπει να χρησιμοποιούν Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ πολύ σύντομα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή και την σκιώδη εισηγήτρια που πήρε ήδη το λόγο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, παρόλο που αν κοιτάξει κανείς με μεγαλύτερη προσοχή την υπόθεση, θα συνειδητοποιήσει ότι εδώ μιλάμε για επιβαρύνσεις, έτσι. οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να βελτιώσουν τα πράγματα στο μέλλον, αλλά είναι προαιρετικές σε όλες οι αλλαγές αυτές, δεν είναι καν υποχρεωτικές. Τα φορτηγά τελικά είναι τα εύκολα θύματα. Κανείς δεν αγαπάει τα φορτηγά, οπότε επιβάλλονται ορισμένα πράγματα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να ε, γίνουν όμως κάποιες συζητήσεις και η εσωτερικοποίηση κάποιων εξωτερικών του εξωτερικού κόστους είναι μια ιδέα που α, είναι ε, που, πρέπει να προωθηθεί. Από την άλλη μεριά το earmarking είναι πολύ σημαντικό για μας. Δηλαδή κάποια κονδύλια να δεσμεύονται για ακά που για κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Από την άλλη μεριά βέβαια αύριο μπορεί να αποφασίσουμε ότι μπορούμε να δούμε ότι χρειάζονται κονδύλια για άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, έχουμε τα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα, έχουμε το Γαλιλαίο και ε, ξέρουμε ότι η συνέχεια του Γαλιλαίου θα κοστίσει. Άρα γιατί δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε... Ε, ε, κάποια κονδύλια από ένα είδος μεταφοράς και να τα χρησιμοποιήσουμε για να συγχρηματοδοτήσουμε αν θέλετε και άλλου είδους πολύ σημαντικά σχέδια που οδηγούν σε ε, πιο ευφυείς μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισεν. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί ελέγξαν πολλά από αυτά που ήθελα να πω. Είναι όντως κρίμα να, που μπαίνουν εδώ μοναχά τα φορτηγά και τίποτε άλλο. Κρίμα. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε παραπάνω πράγματα εδώ. Τέλο πάντων, εύχομαι στον εισηγητή καλή επιτυχία με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Από εκεί και πέρα για το earmarking και τη στοχευμένη αν θέλετε χρησιμοποίηση κονδυλίων, όντω καταλαβαίνω ότι αν προέρχονται από τι οδικέ μεταφορές θα πρέπει να βοηθήσουν τι οδικές μεταφορές. όμω υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι το

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλα πράγματα. Και σε τελευταία ανάλυση και το Υπουργείο Οικονομικών φαντάζομαι και το κοινοβούλιο μας θα πει ότι εδώ τίθεται θέμα ε, εθνικής κυριαρχίας και δεν μπορεί να λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πάνε τα λεφτά μας. Ο επόμενος ομιλητής. Κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Μέχρι τώρα δίνονταν πάρα πολλά κρατικά χρήματα για την δημιουργία κατασκευή καινούριων δρόμων για τις οδικές μεταφορές. Έφτασε και η στιγμή επιτέλους κάποια ε, έσοδα να ξαναγυρίσουν στο, στο κράτος για να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω επενδύσεις. Ε, το, τα φορτηγά δημιουργούν κόστη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα τα εξωτερικά κόστη να, ε, να εσωτερικοποιηθούν και βεβαίως δεν είναι κανένα πρόβλημα ε, τα φορτηγά τα οποία ε, ούτως ή άλλως ε, ζημιώνουν και βλάπτουν το περιβάλλον να κάνουν κάτι για το περιβάλλον πλέον για το όνομα του Θεού από εκεί και πέρα τώρα για το, τη συμφόρηση αυτό δεν είναι καν θέμα δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε για τη συμφόρηση όταν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για το, το περιβάλλον και το θόρυβο και τα λοιπά που προέρχεται από τα διακοπή. Από εκεί και πέρα η συμφόρηση και το earmarking όπως και το earmarking είναι δευτερεύουσα σημασίας. Τώρα, τουλάχιστον ίδια, α, ίδιες συνθήκες και ίδια ίδιοι όροι όπως και για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα για το Euro 5 και Euro 6 τι να σας πω. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν με ενδιαφέρει να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι μολύνουν. Αυτοί που μολύνουν πρέπει να α, ας τους δώσουμε κάποιο κίνητρα ωραία για να προσαρμοστούν. Αυτοί πρέπει όμως να τιμωρηθούν κατά κύριο λόγο για να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Ο κύριος Βαντάλ, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλύτερα να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα παρά ασάφειες. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε τέτοιου είδους λύσεις. Δεύτερον, ως Επιτροπή Μεταφορών εμείς θα πρέπει να διαμορφώσουμε μία θέση και να στείλουμε τον εισηγητή μας σε διαπραγμάτευση. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει ως Επιτροπή εμείς να υιοθετήσουμε μια συγκεκριμένη στάση. Το θέμα αυτό της διαφοροποίησης της τιμής των διοδίων είναι ένα θέμα σημαντικό, θα πρέπει να το λύσουμε, αλλά και επίσης το θέμα της ε, ε διαλειτουργικότητας είναι σημαντικό. Όσον αφορά τις κλάσεις, κυρίως την κλάση 6, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την διαπραγματευτούμε ανάλογα με το κάθε φορτηγό. Τα έσοδα επίση είναι σημαντικό θέμα. Θα πρέπει όμως να διαμορφώσουμε θέση για να μπορέσουμε σιγά σιγά να διαπραγματευτούμε με την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρένερ, η κυρία Κάτσου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πάρα πολύ σύντομη. Εγώ υποστηρίζω την, έκθεση του ΣΑΙΔ διότι έχει μια ελάχιστη αν θέλετε ρεαλιστική συνιστόσα ε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ε, ε, μιλάμε για πράγματα στα οποία έχουν τεράστια συμφέροντα αν θέλετε τα κράτη-μέλη και άρα το Συμβούλιο. Από την άλλη μεριά ξέρουμε πολύ καλά ότι τα διόδια ή μόλις τα ορισμένα αυτοκίνητα α, κάποιων μεγεθών επηρεάζουν, μολύνουν την α, ατμόσφαιρα ε, κάτι πρέπει να γίνει εκεί αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις εναέρες και τις θαλάσσιες μεταφορές και ε, και οι συνερο... σιδηροδρομικές μεταφορές είναι αυτές που πρέπει να ανταγωνιστούν τις οδικές μεταφορές κατά την άποψή μου ίσως θα πρέπει να τονιστούν λίγο παραπάνω σιδηροδρομικές μεταφορές στην έκθεσή του Grazie Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα πολύ λεπτό. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόθεση αύξηση των διοδίων για τις οδικές μεταφορές. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορέσετε να το εφαρμόσετε το σύστημα αυτό. Εγώ συμφωνώ, αλλά μέχρι σήμερα πρέπει να πω ότι βασίζουμε την, τα τέλη ανάλογα με την χρήση. Τώρα προσθέτουμε ένα άλλο κριτήριο. Αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο και αυτοί που ρηπαίνουν περισσότερο. Σωστή και λογική είναι η αρχή, αλλά πώς θα την εφαρμόσουμε στην πράξη. Οι χρήστες τελικά είναι αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν, καθώς και οι αυτοβιομηχανίες. Βεβαίως και θέλουμε να έχουμε λιγότερη ρήπανση στην Ευρώπη, αλλά δεν βάζουμε ούτε ένα ευρώ από την τσέπη μας τι θέλουμε, να πληρώνουν μόνο όσοι περνούν από αυτοκινητοδρόμους, οι, οδηγοί των φορτηγών. Δεν είναι εθνικό το θέμα αυτό, ξεπερνάει τα όρια της κάθε χώρας. Είναι διεθνές το πρόβλημα. Επίσης, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πιο ελκυστικό στα πλαίσια του παραντός συστήματος. Κάτι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε για τις κλάσεις 5 και 6. Αλλά πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Τα κράτη. Πρώτα απ' όλα. Επίσης, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να κανονίσουν, να ρυθμίσουν κατά κάποιο τρόπο τα θέματα της ε, ε διέλευσης. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ε, της Επιτροπής, δεν θέλω να σας πιέσω ούτε να σας περιορίσω το χρόνο, απλώς σας υπενθυμίζω ότι Μακρυμογορήσαμε πολύ για αυτό το θέμα να στη προσεκτικοί. έχει σημασία για μας το θέμα του Δικομισιού. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν προσπαθούμε, όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοί σας, να βάλουμε στη θέση του κατηγορούμενοι πάντα τα φορτηγά. Θέλουμε να κάνουμε κάτι για την Ευρωβουλία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ε, στοιχεία, τα κονδύλια, το κόστος, το κάναμε αυτό με τις εκπομπές αερίων, κάναμε κάτι για τις ενεργοφορίες, κάναμε κάτι και για τις ε, συνδρομικές μεταφορές και τώρα συζητούμε το θέμα με την εναυτιλία. Δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε κανένα. Ούτε καν στους δρόμους, γιατί ξέρουμε ότι οι οδικές μεταφορές είναι το 80% των χερσαίων ε, μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, στα πλαίσια του Λευκής Βίβλου θα δούμε πώς θα ορίσουμε το θέμα αυτό του κόστους για να έχουμε ένα σύστημα πιο βιώσιμο, πιο αηφόρο και να συνεισφέρει όλο αυτό το σύστημα και στην οικονομική ανάπτυξη και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς στόχους που προβλέπεται στα πλαίσια στρατηγικής του 2020. Η έγκριση λοιπόν της οδηγίας πραγματικά πρέπει να σας πω ότι είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αξιοπιστία στις πολιτικές μας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό λαμβάνοντας υπόψη την πραγματιστική προσέγγιση την οποία διαβλέπω εγώ στα πλαίσια των συζητήσεων αυτών. Το Συμβούλιο πρέπει να πω ότι, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι δέχθηκε παρά τις δυσκολίες το θέμα της ε, ε, εσωτικερίδες του κόστους. Μπορέσαμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα μετά από προσπάθειες που κατέβαλε η Βελγική Προεδρία, διότι υπήρχε μια κάποια στασιμότητα στο παρελθόν. Τώρα, για τα θέματα που αναφέρθηκαν, το πιο σημαντικό είναι το earmarking, δηλαδή το θέμα της ε, ε, χορήγησης κάποιων κονδυλίων. Θα πρέπει να είστε πραγματιστικοί, να μην μπλοκάρουμε τα πράγματα. Πώς σας λέω θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. το επαναλαμβάνω. Το Συμβούλιο δεν έχει πολύ μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι όπως είπε και ο συγητή, υπάρχει περιθώριο μιας κάποια πρόοδο στον τομέα αυτό. Και θα πρέπει να διορθωθεί το τεχνικό σφάλμα το οποίο υπήρχε στην κοινή θέση όπου ε, δεν ληφθεί υπόψη το καλό αποτέλεσμα και η συμφωνία στην οποία είχαμε καταλήξει για την αναθεώρηση των τελών. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και κάποιος τρόπος να γίνουν πιο ορατά τα πάντα όσον αφορά τα έσοδα τα οποία ε, έχουν αυτοί που εισπράττουν τα τέλη και πώς τα χρησιμοποιούν. Θα πρέπει να βρεθεί και κάποια λύση για το θέμα αυτό της, ε, των ε, ανταλογών Καυτερίνωση στα πράσινα της σχετικής οδηγίας και να δούμε τι γίνεται με τα θέματα μείωσης της ρήπανσης. Θα μπορούσε αυτό το θέμα λοιπόν του Market, της ε, δέσμευσης κάποιων κονδυλίων για αυτά τα θέματα να προσπαθήσει να τα περάσει το Κοινοβούλιο στην ε, συμφωνία. Τώρα, το θέμα των διαφοροποίησης των διοντίων στις ώρες εχμής. Το παρόν κείμενο του Συμβουλίου προβλέπει ανάλογα με την ώρα διέλευσης κάποιο διαφορεμένο κόστος κατά το όριο σε ποσοστό 175% πάνω από το κανονικό ποσό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και επί του παρόντος, αλλά με πολύ μικρότερο ε, περιθώριο αυτή. Αυτή η καινοτομία αυξάνει περιθώρια κατά σημαντικό τρόπο. Πρώτα απ' όλα διότι η διαφοροποίηση είναι πιο μεγάλη από το μέσον όρο και όχι από το ελάχιστο, έτσι όπως προβλέπετε στο νομοθετικό κείμενο. Είμαστε λοιπόν πολύ κοντά στις προτάσεις και στις ε, τροπολογίες που κατέθεσε πρώτη ανάγκη στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Κάναμε κάποιες ασκήσεις προσωμείωσης και είδαμε ότι το 195% σχέση με το μέσον όρο σχεδόν καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα ε, στο οποίο κατέληγε και η προηγούμενη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή στο ελάχιστο όριο αύξηση του κατά 500%. Η Κομισιόν λοιπόν δεν θέλει να υπάρχει μεγάλη αλλαγή στο πάνω Αυτό το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε είναι η διάρκεια, η ημερήσια χρονική διάρκεια αυτού του τέλους των ωρών ε, εχμήν. Πέντε ώρες, λέει το Συμβούλιο και μπορεί να καταθέσει ως τροπολογίες θέλει επί αυτού του χρονικού διαστήματος το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, η κλάση 6 και η εξαίρεση. Στην κοινή θέση προβλεπόταν τρία χρόνια. Άρα η κλάση 6 αν θέλετε, θα επωφεληθεί από ένα μπόνους, από ένα κίνητρο, ακόμη ένα χρόνο. Εάν μειωθεί ο χρόνος μεταφοράς, τα θα πρέπει επίσης να μειωθεί και η περίοδος εξαίρεσης της κλάσης 6. Και δύο τελικά σχόλια, στόχος και δύο λειτουργικότητα. Ο στόχος είναι να καλυφθούν τα φορτηγά 3,5 με 5 τόνους. Εδώ πρέπει να πω ότι δεν συμφωνούμε με την κοινή θέση που διαμορφώθηκε. Δεν είμαστε διαδογματικοί τόσο αφορά ποια φορτηγά θα πρέπει να καλύπτουν, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ο κανόνας ο ίδιος για όλα τα κράτη-μέλη, διότι δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη να εξαιρέσουν ανάλογα με το τον κάποια φορτηγά. Και νομίζω ότι θα μας βοηθούσε να είμαστε πιο ορθολογιστικοί. Τώρα, Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, σας διαβεβαιώνω ότι εμείς από τη μεριά μας αυτό το θέμα το προσέχουμε ιδιαίτερα. Υπάρχει το, για το 2013 η πρόβλεψη να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή η οδηγία διαλειτουργικότητας και βεβαίως είναι, έχει ευθυγραμμιστεί το σύστημα αυτό της Ευρωβουλίας σε αυτό το θέμα. Διευκρίνηση κύριε Μπρόνμπουρ, αν θέλετε να είστε πάρα πολύ γρήγορος παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Απλώς διερωτώ με μήπως ε, εάν χρειαστεί μπορεί να μου απαντήσει και γραπτά. Ε, δηλαδή υπάρχει κάποια έκθεση αντικτύπου, ε, μια έρευνα για το ποιες είναι οι συνέπειες. Δεν θέλω να ξαναδείξω τη συζήτηση τώρα. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Παρόμοια ερώτηση. Πρόεδρε, εγώ ε, έθεσα μία ερώτηση στην Κομισιό και δεν πήρα απάντηση. Το κόστος εισαγωγής του, του όλου συστήματος. Έχετε συμφωνήσει για το ποιο... ποιο τι θα πληρωθεί από ποιον. Λοιπόν, ετέθησαν δύο ερωτήσεις. Μπορεί να απαντήσετε ναι ή όχι, να τελειώνουμε. Ναι. Έχουμε, έχουμε κάνει μια αξιολόγηση αντικτύπου, ενδελεχέστατη θα έλεγα, και όλες αυτές οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Εισηγητή, δύο λεπτά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τον πιο γρήγορα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον και για τα σχόλια τα οποία έκαναν. Πολλές ερωτήσεις απαντήθηκαν από την Κομισιόν, κυρίως όσον αφορά ε, το, τη διακύμανση, αν θέλετε, ε, του τέλους ε, προφανώς αυτή η διακύμανση θα πρέπει να προσαρμοστεί για κάποιο συγκεκριμένο διάδρομο, έτσι ώστε όλα, ανά διάδρομο μάλλον, έτσι ώστε τα, ε, όλα τα οχήματα να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο το σύστημα. Όσον αφορά το earmarking, είπα ήδη και το είπα και στο Συμβούλιο, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για μας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια, θα πρέπει να γίνονται οι εκθέσει κανονικά και ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στην νομοθεσία μας. Και μπορούμε βέβαια να ε, εμπνευστούμε από την νομοθεσία για την ε, εμπορία των εκπομπών. Τώρα, η άποψη του Κοινοβουλίου είναι ότι μπορούμε να συνδυάσουμε κάποια πράγματα εδώ αναφερόμαστε ε, στο εξωτερικό κόστος ή το earmark. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα περισσότερο λιπογόνα οχήματα. Εκεί μπορούμε να συνδυάσουμε το markup και, κάποια, και να το συνδυάσουμε και με το εξωτερικό κόστος. Τώρα για τα άλλα οχήματα 5, 6, 4, 5 και 6 δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση. Όμως θέλουμε και σε αυτό και σε αυτή την κατηγορία να δώσουμε ένα κίνητρο για να αποσύρουν, τα, να ανανεώσουν το πάρκο. Εάν δούμε το κείμενο το οποίο διαπραγματευτήκαμε το 2006, είχαμε πει έπρεπε μέχρι το 2012 να έχουμε 305, 305 τόνους. Αυτός ήταν ένας τρόπος να παρακάμψουμε αυτή την ε, υποχρέωση, αλλά ε, θα πρέπει για να γίνει κάτι τέτοιο να έχουμε συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε στο Συμβούλιο, ότι δεν μπορούμε να τους δώσουμε μια επιταγή εν λευκό. Τώρα, υπάρχει μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και σαν εισηγητή μπορώ να δεσμευτώ να έχουμε ειλικρινείς διαπραγματεύσεις, όμως για να γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να, να καταλήξει η Επιτροπή σε κάποια απόφαση, κάποια άποψη και θα πρέπει να επωφεληθούμε από, όσο το περισσότερο από τον λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Επομένως, αυτό το οποίο προτείνω είναι να δούμε εάν υπάρχει περιθώριο για συμβιβαστική, ε, συμβαστικές λύσεις, ε, εισηγητής, ε, κτλ. Για, και να προχωρήσουμε. Τώρα, η ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, μεταφορών μπορεί να γίνει αφού έχουμε άτυπες συζητήσεις με το Συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικειωθούμε περισσότερο με τα γεγονότα και θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, ε, ε, να δούμε τις απόψεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων και θέλω όμως μια εντολή για να ξεκινήσω, γιατί ούτως ή άλλως θα υπάρξει μετά ένας επίσημος τρίλογος. Όμως για να ξεκινήσω ο επίσημος τρίλογος πρέπει να έχει το κοινοβούλιο άποψη. Δηλαδή θα πρέπει να ψηφίσει η Επιτροπή και μέσα στα πλαίσια εκείνου του τριλόγου θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ή και να καταλήξουμε ενδεχόμενα. Και αν δεν υπάρχει ε, φως για συμφωνία μπορούμε να περάσουμε σε δεύτερη ανάγνωση. Πρόεδρος, συμφωνείτε ο εισηγητής να ξεκινήσει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις για να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Και αφού οι σκιώδεις εισηγητέ και ο εισηγητή καταλήξουν σε κάποια απόφαση, σε κάποια άποψη, να επανέλθουν στην Επιτροπή, να την επισημοποιήσουμε αυτή την, απόφαση, την και μετά να ξεκινήσει ο επίσημος τρίλογος. Και αυτά, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι, ε, γίνεται κατά εξαίρεση, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Το φοβόμουνα, το φοβόμουνα. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε συζητήσεις για διαδικασία. Απλώς να τονίσω ότι για πολλές πολιτικές ομάδες υπάρχουν ερωτηματικά, διότι είναι καινούργια το Κοινοβούλιο. Επομένως δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία τώρα, δεν λέω. Αλλά μήπως θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε κάπως την διαδικασία ε, με την υποβολή του σχεδίου έκθεσης. Ξέρουμε ποια είναι τα θέματα ε, ε, και ξέρουμε και τις αναλλακτικές. Θέλουμε μια επιταχυμένη διαδικασία. Πρόεδρος. Με την ε, σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής ε, θα πρέπει ο εισηγητής ε, να συζητήσει με τους σκιώδεις και να συντάξουν μια έκθεση η οποία θα υποβληθεί στην Επιτροπή όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Κύριε Στέρξ, σας κατάλαβα καλά για την, ποια θα είναι διαδικασία. Ο Σαΐντ θα συνεδριάσει μαζί μας, θα υποβάλουμε μια πρόταση στην Επιτροπή και μετά προχωράμε στον Τρίλογο. Πολύ ωραία. Δεν μπορεί να ξεκινήσουμε τρίλογο εάν δεν έχει διαμορφωθεί άποψη της Επιτροπής. Πρέπει να έχουμε τη θέση της Επιτροπής για να ξεκινήσει ο τρίλογος. Ωραία λέει ο κύριος Αλκαντράουι. Το ξέχασα. Θα πρέπει να συζητήσουμε την, ε, μια, τις συμβιβασμού ε, μέσα σε έναν επίσημο βέβαια πλαίσιο. Κάτι το οποίο συμφωνήσαμε και τον ε, Δεκέμβριο στην Επιτροπή μας. Whatever informal discussions you want to have as rapporteur in consultation with your shadows with the council Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, μια συζήτηση με τους σκιώδεις. Ε, από εκεί και πέρα οι επαφές με το Συμβούλιο είναι δική δικό σας θέμα αν θέλετε, ανεπίσημα. Όμως τρίλογο δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε αν δεν διαμορφωθεί και δεν παγιωθεί η άποψη της ε, Επιτροπής μας. Όμως αυτό το οποίο, ε, για το οποίο μπορούμε να σας, αυτό που μπορούμε να σας ε, εμπιστευτούμε συγγνώμη, είναι να διαμορφώσετε εσείς και οι σκιώδεις μία θέση και να τη συζητήσετε με το Συμβούλιο ενδεχόμενα. Και γίνεται αυτή η διαδικασία ακριβώς επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ήδη από την πρώτη ανάγνωση άλλαξε το κοινοβούλιο, όπως το είπαν και οι συνάδελφοι. Γι' αυτό θα πρέπει οι σκιώδεις και ο εισηγητής να, να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, να διαπραγματευτούν ε, κάποια πράγματα με το Συμβούλιο, γιατί κάποια πράγματα μπορούν να διαπραγματευτούν, κάποια όχι. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα, δική σας απόφαση. Στη διακριτική σας ευχαίρεια είναι. Και μετά θα, θα έρθετε στην Επιτροπή. Πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ε, ε, ο εισηγητής είναι ελεύθερος να συναντηθεί με τους σκιώδες, με τους συντονιστές και μετά από αυτή τη συνάντηση να διαπιστώσει τι πρέπει να κάνουμε διότι όπως ελέγχθη χρειαζόμαστε μεγαλύτερες πλειοψηφίες αν πρόκειται να διεκδικήσουμε και να επιμείνουμε σε κάτι έναντι του Συμβουλίου. Ε? αν δεν γίνει κάτι τέτοιο τότε να καθίσουμε σπίτι μας καλύτερα. Πρόεδρος, ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Οι, οι και οι σκιώδεις πρέπει να κάνουν δουλειά τους τελικά, ε, για να είμαι τελείως χοντροκομμένος. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την, Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, το οποίο είναι η δική μου έκθεση. Λοιπόν, εγκαταλείψτε το κτίριο σαν γρήγορα. International Air Agreement διεθνείς συμφωνίες για την ενέργεια κυκλοφορία ε, μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Όταν ζήτησα όσοι θέλουν ε, να καθυστερήσουν τη συνεδρίες να το κάνουν έξω από την αίθουσα, σας παρακαλώ. of includes the Council and the Commission especially. Λοιπόν, όσοι θέλουν να συνεδριάσουν, ε, ιδίω ε, το Συμβούλιο ή την Κομισιό, α το κάνουν έξω. Εκείνοι δεν μας επιτρέπουν στο Συμβούλιο, δεν μας επιτρέπει να ε, συνεδριάζουμε στο εσωτερικό των δικών του συνεδριάσεων, άρα ούτε και εγώ θα του το επιτρέψω. Μπορείτε να καταλήψετε την αίθουσα σας παρακαλώ για να συνεχίσουμε. Όπως συζητήσαμε τον Οκτώβριο, πρόκειται για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που αντικατοπτρίζει τις νέες συμφωνίες τις, μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, εκεί που απαιτείται η σύμφωνη γνώμη, η συνένεση του Κοινοβουλίου πριν ολοκληρωθεί μια διεθνής συμφωνία. Υπάρχουν τα διάφορα είδη συμφωνιών και πριν πω αυτό, ε, είμαστε η έκθεση χωρίζεται σε τρία τμήματα σε δύο τμήματα. Το ένα είναι η συμφωνία αυτή καθεαυτή και μετά είναι τα το περιεχόμενο της συμφωνίας και μετά η παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά το περιεχόμενο δεν πρόκειται να επαναλάβω, αυτά που είπα προηγουμένω ε, για τις ε, ε, συμφωνίες. Οι συμφωνίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα και στους επιβάτες και σε αεροπορικές εταιρείε, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται οι υπηρεσίε και περιορίζεται το κόστος μέσα στα πλαίσια ενός υγιούς ανταγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη και το κοινωνικό κόστος. Επίσης, ε, εξασφαλίζουν μια νομική σαφήνεια ε, που όλοι οι δικηγόροι θέλουν να έχουν. Το σχέδιο έκθεσης τώρα ε, αναφέρει διάφορα κριτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση μιας συμφωνίας. Μιλάμε για την ισορροπημένη πρόσβαση στην αγορά, τήρηση υψηλών ε, περιβαλλοντολογικών ε, ε, συνθήκων, εξασφάλιση των, της προστασίας των δεδομένων, δικαιώματα των επιβατών. Επειδή δεν έχουμε πολύ, χρόνο, χώρο στη διάθεσή μας για αυτές τις εκθέσεις, πάρα πολλά θέματα αναφέρονται ιδιαίτερα συνοπτικά διότι ούτως ή άλλως σε μια έκθεση πρωτοβουλίας έχουμε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όσον αφορά τις επεξηγηματικές, ε, ε, την εισαγωγή τέλος πάντων, θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση για όλες τις συμφωνίες. Ταυτόχρονα όμως δεν λέει κανείς ότι κάθε, συνθήκη πρέπει να σέβεται ένα κατάλογο θεμάτων τα οποία πρέπει να πληρούνται για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η επιμέρους συμφωνίες, σύμφωνα με το οποίο μάλλον ε, πρέπει μπορούν να κριθούν, να αξιολογηθούν οι επιμέρους συμφωνίες και οι επιμέρους εισηγητές να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Τη ζήτηση που είχαμε τον Οκτώβριο καταλήξαμε σε μία ε, συμφωνία ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί τις συμφωνίες, ε, τις διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις όσο αυτές εξελίσσονται και να μην περιμένει το τέλος της ε, επίτευξης συμφωνίας. Συζητήσαμε με τον κύριο Κάλλας ε, για να δούμε πώς οι διατάξεις ε, της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαίσιο ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν θα πρέπει να αναφερθούν σε περιπτώσεις διεθνούς συμφωνίας για τις μεταφορές. Στην επιστολή που μου έστειλε στις 19 Ιανουαρίου επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η, η Κομισιόν, οι υπηρεσίες της Κομισιόν είναι στην διάθεσή μας να μας ενημερώνουν για τις διαπραγματεύσεις όσο εξελίσσονται και, στο παράρτη, και, και πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα 3 τη ε, της Συμφωνίας Πλαίσιο ε, θα παρουσιάζονται, θα είναι στη διάθεσή μας. Όπως σας είπα, ε, υπάρχουν ε, όρια όσον αφορά την, ε, το μέγεθος αυτής της ε, ε, έκθεσης πρωτοβουλίας. Επομένως ενημερώνω και προειδοποιώ τους σκιώδεις συζητητές ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θίγονται με, πολύ πιο συνοπτικά από ό,τι θα θέλανε και εκείνοι και εγώ. Αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια έκθεση η οποία θα εξασφαλίσει μια ευρύτερη συμφωνία και που θα καθορίσει ε, τα πλαίσια ε, μέσα στα οποία οι εισηγητές του Κοινοβουλίου θα μπορούν να εργαστούν ε, για αυτές τις τόσο σημαντικές συμφωνίες στον τομέα των εναέριων των αεροπορικών μεταφορών. Λοιπόν, εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε μελέτης διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση η οποία ρίζει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και άρα δεν υπάρχουν ερωτήσεις αλλά ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες συστάσεις αν θέλετε τον Οκτώβριο ήδη είπαμε ότι θα πρέπει από την αρχή ε, να συμμετέχει σε οποιασδήποτε συζητήσει του Κοινοβούλιο γιατί είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένουμε σε αυτό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Στις όλες... Ε, στις, διμερείς συμφωνίες ας πούμε που έγιναν με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τα λοιπά είδαμε ότι ε, υπήρξαν και ότι υπή, καλύπτεται η περίπτωση σε μονομερούς καταγγελίες και τα λοιπά. Και γι' αυτό λοιπόν ε, στις εναέριες μεταφορές μια και ε, η τεχνολογία τρέχει και τα πράγματα αλλάζουν ιδιαίτερα μετά από, την, ε, από το φοβερό την τραγουδία στο αεροδρόμιο της Μόσχας θα πρέπει να έχουμε και εδώ κάποιες ρήτρες αν θέλετε ευελιξίας ο, θα πρέπει και όλες αυτές και οι συμφωνίες που υπάρχουν να μπορούν να τροποποιηθούν, να προσαρμοστούν σε μια ρευστή εξωτερική κατάσταση. Και, αυτό λοιπόν ήθελα να πω. Ήδη από την αρχή της διαπραγμάτευσης να λαμβάνει μέρος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις συζητήσεις και να υπάρχει μια κάποια ληξία λόγω του ρευστού του διεθνούς περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εσύ, Νομίζω ότι πολύ καλή ήταν η παρουσίαση του θέματος. Νομίζω ότι μπορούμε να σας υποστηρίξουμε και πρέπει να σας πω ότι για μας το θέμα αυτό το σενάριας ε, κυκλοφορίας και της ελευθερίας όταν υπάρχουν σωστές συμφωνίες ήταν ένα για μας θέμα προτεραιότητας. Θα πρέπει το κόστος να είναι ακόμη για τις τρεις χώρες το ίδιο. Το ίδιο για όλους. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Επίσης, το λέγω αυτό για να μην υπάρχει αθέμητος συναγωνισμό. Μιλήσατε επίση για τι συμφωνίες που έχουμε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και ΕΕ. Πρέπει να πω ότι έχουμε την κατάλληλη βάση για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Ε, πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξέρει περί τίνος πρόκειται, διότι εκεί παίρνονται οι αποφάσει και εκεί προετοιμάζεται το μέλλον και ό,τι μα επηρεάζει θα πρέπει να το γνωρίζουμε. οι ενδιαφερόμενοι, οι διάφοροι φορείς, οι επιχειρήσεις είναι παρόντες. Γιατί όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν όχι γιατί να μην λαμβάνουμε εκ των προτέρων την, την ημερήσια διάταξη και εκ των υστέρων τα πρακτικά για να ξέρουμε τι ακριβώς συζητείτε. Επίσης πιστεύω ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι τα δικαιώματα των επιβατών, των χρηστών των αεροπορικών εταιρείων. Μετά από τα προβλήματα που είχαμε πέρσι με τη στάχτη στην Ιλανδία, είδαμε τι προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν. Και είδαμε τι κανόνες εφαρμόζονταν για αυτούς οι οποίοι ξεκινούσαν από την Ευρώπη με μία ευρωπαϊκή εταιρεία, αλλά τι δικαιώματα έχουν οι επιβάτες τρίτων χωρών ή αυτοί που απλώς περνούσαν από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει τα δικαιώματα των επιβατών τουλάχιστον στην Ευρώπη να εφαρμόζονται σωστά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ, κύριε Λακαντράγκη, κοιτάξτε την παράγραφο. Κοιτάξτε, αυτό το τελευταίο ήθελα να πω κι εγώ, ότι τα δικαιώματα των ε, επιβατών πρέπει να προστατεύονται, αλλά υπάρχει παράγραφος 6. Το πρόσκησε αυτό ο εισηγητής. Τέλος πάντων, είναι εδώ εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι είχαμε κάνει και μια ε, έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας το 2005 και είχαμε πει ότι πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα. Τότε παρακαλούσαμε. Τώρα όμως η, ε, συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει κάποια δικαιώματα. Θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι. Παρακαλούσαμε παλιά για πληροφορίες. Τώρα είναι υποχρεωτικό να μας δίνονται οι πληροφορίες αυτές και αυτές πρέπει να τις απαιτήσουμε. Τώρα, για τις ε, ε, συμφωνίες με την Κίνα και την Ινδία. Αυτό που λέγεται είναι σωστό. Η Κομισιόν έχει την ε, διαπραγματευτική εντολή, αλλά πολύ σημαντικό να τονίσουμε είναι επίσης ότι θα πρέπει να υφίστανται παρόμοια πλαίσια παραδείγματος χάρη κρατικών ενισχύσεων σε όλες τις χώρες για να μπορούν να προχωρήσουν οι συμφωνίες αυτές. Για να ξέρει κανείς τη συμφωνία για να, να είναι δίκαιες οι συμφωνίες. Επίσης, εκείνο που είναι σημαντικό για, μα, μένα και αναφέρεται πάλι στην παράγραφο 6 η, σε σχέση με την αξιολόγηση των συμφωνιών είναι το εξής. Η, βεβαίως είναι, ε, αναφέρονται εδώ ε, σε σχέση με την τρομο, τρομοκρατία ε, και τους σκάνερς και τα νούμερα για τους επιβάτες και τα λοιπά ε, πού συλλέγονται όλα αυτά τα στοιχεία και τι γίνεται με τα προσωπικά στοιχεία τα μεταξύ αυτών που συλλέγονται ή θα πρέπει να ξέρουν να υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές για να ξέρουμε ακριβώς τι συμφωνούμε για να ξέρουμε αν είμαστε υπέρ ή κατά μια συμφωνίας για να υπάρχει διαφάνεια στη συμφωνία διότι διαφορετικά εγκρίνουμε ή απορρίπτουμε μη διαφανή πράγματα πράγματα για τα οποία δεν ξέρουμε τίποτε αν λοιπόν μου πείτε ότι πράγματι θα υπάρχει διαφάνεια και θα ξέρουμε που ε, και πώς συλλέγονται τα στοιχεία αυτά τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα με την έκθεση ευχαριστώ πολύ κυρία Φώστερ ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ για την ε, περιστατωμένη σας έκθεση. Το, κάποιες παρατηρήσεις γενικής φύσεως πρώτα-πρώτα. Έχετε δίκιο. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση την περασμένη φορά και αναφέρθηκαν πολλά θέματα από, από μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο που θα πρέπει να παίξει το Κοινοβούλιο. Εγώ συνεχίζω να επιμένω ότι ο πως ε, δέχτηκε και ε, ο Επίτροπος τελικά ε, ότι επιμένω ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις βεβαίως δεν είμαστε καλοί διαπραγματευτές εμείς ε, δεν, θα πρέπει να αναλάβουμε τον ρόλο του διαπραγματευτή αλλά τέλος πάντων διατηρώ τη θέση μου από αυτού ένα-δυο ακόμη παρατηρήσεις για τα 6 και 7 για το PNR και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνονται όμως σε παραρτήματα ουσιαστικά των ε, συμφωνιών. Δεν περιλαμβάνονται στο σώμα της ε, συμφωνίας. Χρειάζεται να τα αναφέρουμε εδώ αυτά ή όχι. Δεν ξέρω. Πείτε μου. Μία παρατήρηση αυτή, δεύτερη. Παράγραφος 10. Εκεί Λέγεται ότι η Κομισιόν χρησιμοποιεί ουσιαστικά τις συμφωνίες αυτές σαν μοχλό για να προωθήσει ε, εργατικά στάνταρς και πρότυπα. Ε, δεν είναι σωστό αυτό και στη δεύτερη φάση, όταν συμφωνήθηκε αν θέλετε η δεύτερη φάση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ΕΕ, αναφέρθηκαν κάποια σχετικά θέματα αλλά μπήκαν χώρια και πολύ συγκεκριμένα. Δεν νομίζω ότι ε, μπορούμε μέσα των συμφωνιών αυτών να επηρεάσουμε τις τρίτες χώρες για το τι θα κάνουν στην αγορά εργασίας τους ε, υπάρχουν και κάποια όρια τέλο πάντων. Ε, αυτά, θέλω, μπορεί και να μην κατάλαβα καλά την παράγραφο 10 και ένα τελικό θέμα να μας ενημερώσει η Κομισιόν γιατί ένα από τα βασικά θέματα που αναφέρονται εδώ και δικαίω το είπατε πρόεδρε είναι ότι θέλουμε ε, τελείως φιλελεύθερες συμφωνίες δεν είμαστε υπέρ του προστατευτισμού και ο αγώνας αυτός δόθηκε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέρμα έχουμε συμφωνήσει από αυτού. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν τι γίνεται με τη συμφωνία με την Αυστραλία. Εξ οσου γνωριζω γνωρίζω υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, ένα ίσως και παραπάνω, που παίζουν καθυστερητικές τακτικές. Αλλά η, Αυστρά, η συμφωνία με την Αυστραλία είναι μια από τις πιο σημαντικές που θέλουμε να συνάψουμε. Λοιπόν, για πείτε μας μερικά πράγματα, ακόμη περισσότερο αν υπάρχει θέμα εμπιστευτικότητας και απορρίπτου, απορρίπτου εδώ. Εμείς πρέπει να ενημερωθούμε ε, ευχαριστούμε τελειώνοντας πρόεδρε για την έκθεση. Θα την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει το λόγο, κύριος Κόλιτσεκ. Κύριε Κόλιτσεκ, συγγνώμη, δεν σας είδα. Ε, δεν είμαι και πολύ μεγάλος όμως, γι' αυτό δεν με βλέπετε πρόεδρε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας η οποία κατάφερε ό,τι ήταν δυνατό να καταφέρει. Όπως είπε και η τελευταία μιλήτρια, θα ήθελα να τονίσω και εγώ τη σημασία της παραγράφου 10. Αν λέγονται εκεί πολύ σημαντικά πράγματα και Θα πρέπει να νόμισουμε ιδιαίτερα για να, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει, να γίνεται κοινωνικό τάμπι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας που είναι μια πολύ σαφής βάση εργασίας βάσει της οποίας το Κοινοβούλιο θα ασκήσει το ρόλο του στα πλαίσια της νέας συνθήκης Λισαβόνα. Στα πλαίσια των ε, συμφωνιών για την ε, εναέρεια κυκλοφορία μουτά της μουτάντης, αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και άλλες, συμφωνίες, και άλλες συμφωνίες στον τομέα των μεταφορών. Κάνατε μία διαφοροποίηση πολύ οξυδερκή, σωστή, μεταξύ των ε, τριών συμφωνιών για τις ενέργειες ε, μεταφορές και τους τρεις ε, διαφορετικούς στόχους, οριζόντιες συμφωνίες, σφαιρικές συμφωνίες με τις οποίες θέλουμε να φιλελευθερωποιήσουμε την πρόσβαση στην αγορά δίδοντας συγχρόνως και εγγυήσει για την σύγκληση των νομοθεσιών, δεδομένου ότι θέλουμε όλοι οι φορείς να έχουν σωστές συνθήκες άσκησης του ανταγωνισμού. Αναφέρατε συμφωνίες ασφαλείας που είναι απαραίτητες όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας στις εναέριες, στην εναέρια κυκλοφορία, αλλά συγχρόνως να προωθήσουμε και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποίησης εξοπλισμών και αεροσκαφών ώστε να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε την κατασπατάληση πόρων στις ε, ε, βιομηχανία του κλάδου. Στην αιτιολογική σας έκθεση βλέπω να υπάρχει συνένεση όσον αφορά τις συμφωνίες αυτές. Και όπως υπογραμμίζεται, Οι συμφωνίες αυτές δεν γίνονται για να συνάψουμε συμφωνίες. Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη ευχαρίστηση αν δεν είναι ίσως κελισμένες ε, οι συμφωνίες και δεν θέλουμε να τις επιτύχουμε με οποιοδήποτε τίμημα. Και εδώ νομίζω ότι μπορώ να χαιρετήσω την ιδέα σας να θεσπίσετε κριτήρια, να θεσπίσουμε μάλλον κριτήρια που θα μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε απολύτως ποια είναι η προστέμενη αξία κάθε συμφωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε, να λέμε τα ίδια πράγματα, να είμαστε σταθεροί και ξέρουμε ότι παρόλα αυτά κάθε συμφωνία είναι ιδιαίτερη. Οι στόχοι βεβαίως είναι κάθε φορά συγκεκριμένη, λαμβάνοντας υπόψη και με ποια χώρα διαπραγματευόμαστε. Το θέμα επίσης του ελέγχου και της ιδιοκτησίας είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε αν θέλετε τα ίδια αποτελέσματα όταν διαπραγματευόμαστε με τον Καναδά ή με τις ΗΠΑ όταν διαπραγματευόμαστε με τις αναδυόμενες χώρες Φερρυπίν, νομίζω ότι θα ήταν αυτά πάτη να πιστέψουμε ότι με την ε, διαπραγμάτευση κάποιων ε, κανόνων όσον αφορά να υφερεί την προστασία του περιβάλλοντος θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με τα οποία έχουμε και με άλλους διεθνείς ε, πρωταγωνιστές της των εναερίων μεταφορών. Ούτως ή άλλως, όλες οι συμφωνίες θα πρέπει να έχουν ως στόχο την υλοποίηση των στόχων των δικών μας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, δικαιώματα επιβατών, προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε εμείς με όλα αυτά τις ε, πολιτικές, οι οποίες επί τούτης θα πρέπει και ανάλογα την περίπτωση να εφαρμόσει κάθε Τώρα, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, που είναι αυτό της προστασίας της, ε, των προσωπικών δεδομένων. Με τέτοιου είδους συμφωνίες πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι δεν κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να βλάψει την, ε, τους κανόνες που θέλουμε να ισχύουν για την προστασία της ελληνικής ζωής του κατανάλου στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή, βεβαίως, και εσείς θα πρέπει να κρίνετε ποια είναι τα ωφέλη τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε από μια συμφωνία την οποία θέλουμε να συνάψουμε γρήγορα ή να καθυστερήσουμε εάν θέλουμε, εάν πολλές φορές είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι και δεν καταλήγουμε πουθενά. Θα πρέπει λοιπόν ώρες-ώρες να βλέπουμε και κατά περίπτωση πως έχουν τα πράγματα. Πράγμα που δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμόζουμε τα πάντα ανάλογα με την περίπτωση, αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο οι διάφορες συμφωνίες ε, είναι χρήσιμες ποιος είναι ο στόχος τους και θα πρέπει, όπως είπα, για να προχωρήσουμε θετικά για να συνεχίσουμε το διάλογο, να δούμε ποιος είναι και ο θεσμικός διάλογος ο οποίος έχει αρχίσει και μεταξύ ημών και του Επιτρόπου για να δούμε πώς θα συνεργαστούμε και πώς θα ανταλλάξουμε πληροφορίες και εμείς βεβαίως στην Κομισιό όλες τις χρήσιμες πληροφορίες θα σας τις διαβιβάσουμε στα πλαίσια των δυνατήτων για να προχωρήσουμε. Υπάρχει λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο, η Κομισιόν θα το σεβαστεί και είμαστε έτοιμοι από τώρα όταν και εσείς επιθυμείτε και τηρώντας τους κανόνες του απορρίτου πάντα να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας για να σας ε, διηγούμεθα πώς έχουν τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις. Ακόμη και με την Αυστραλία. Κυρία Φώστερ, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή δημοσίω να σας πω που βρισκόμαστε, αλλά εάν θέλετε είμαι διατεθειμένος όταν τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες απορρίτου να σας ενημερώσω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς να απαντήσω εν συντομία. Όπως σας είπα και στην αρχή που παρουσίασα την έκθεση, ο περιορισμός του αριθμού των λέξεων σημαίνει ότι δεν μπορούσα να αναπτύξω κάποια πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τους συναδέλφους. Η παράγραφος 7 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρίτου. Όντως καταλαβαίνω ότι ε, είναι λίγο ξερή η διατύπωση, όμως έπρεπε να τα συμπεριλάβω, ε, δεν μπορούσα να πω παραπάνω. Όπως επίσης ε, για τα δικαιώματα των επιβατών. Δεν μπορούσα να πω σε λεπτομέρειες. Απλώς ήθελα να τονίσω την ε, υποχρέωση να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των ε, επιβατών. Και να τονίσω ότι μιλάμε για ε, κατευθυντήριες γραμμές που δίνουμε στους εισηγητές όταν εξετάζουν κάποιες συμφωνίες. Οι συμφωνίες είναι διαφορετικές. Κάθε μία είναι ξεχωριστή. Η κυρία Φώστερ έθιξε το θέμα των, του διεθνούς, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και, τα, και γι... Εγώ θεώρησα ότι ήμουν υποχρεωμένος να το συμπεριλάβω αυτό, διότι ε, είναι μια συμφωνία του Κοινοβουλίου, είναι επίσημη άποψη του Κοινοβουλίου. Γιατί είναι ένα θέμα που θέλει να συμπεριλάβει το Κοινοβούλιο στις διάφορες συμφωνίες. Γι' αυτό ήθελα και εγώ να το θίξω. Κατανοώ ότι Κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν. Εγώ απλώς σας εξηγώ γιατί το συμπεριέλαβα, γιατί ακριβώς είναι επίσημη άποψη του Κοινοβουλίου και θέλω να το συμπεριλάβω. Επομένως, συνάδελφοι, η 8 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας είναι 15 Μαρτίου και μετά η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα λάβει χώρο τον Μάιο και ελπίζω ότι θα υπάρχει ένα πλαίσιο έτοιμο τέλος πάντων. Λοιπόν, 8 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου η Επιτροπή μας, η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εδώ ολοκληρώνεται το πρωινό μας πρόγραμμα. Τελειώσαμε λίγο νωρίτερα, το οποίο σας πίεσα λιγάκι, θα μπορούσα να είμαι πιο χαλαρό στο χρόνο που σα ε, έδωσα για την ε, Ευρωβινιέτα. Ε, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στις 3 για την ανταλλαγή απόψεων με την Ουγγρική Προεδρία. Καλό σας μεσημέρι.